Ε, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε σχεδόν πληρότητα, λέει ο πρόεδρος. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης στο σχέδιο κυκλοφόρησης στις 4 Δεκεμβρίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίθηκε. Ανακοινώσει. Σας καλωσορίζω καταρχάς στην κοινή συνεδρία Συνομικής Επιτροπής και Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων Θα έρθει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρο, ο κύριο Φαουρέκη στο στον δρόμο. Ο κύριο Κορμπέτ δεν μπορεί να είναι παρόν συνεισηγητή μου σε ένα θέμα τη ημερήσια διάταξη. Έχει ανηλυμένε υποχρεώσει. Κατά την ανταλλαγή απόψεων πάντω θα αναγνωστεί μήνυμά του γραπτό. Σημείο 3. ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας, της νομοθεσίας. Και ως εισηγητής έχω να σας πω τα εξή. Η Γιούρη και η Αύκο, όπως ξέρετε, έχουν ε, εγκαθιδρύσει ομάδα εργασίας, της οποίας το έργο έχει, σχεδόν, έχει πλέον ολοκληρωθεί, με κύρια ευρήματα με κύρια βάση εργασία στα ευρήματα της έκθεσης των δύο συνεισηγητών. Η έκθεση στόχο έχουμε να περιλαμβάνει τα εξής. Έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο περιλάβει. Πρώτον, το στόχο της υψηλής ποιότητας της καταρτιζόμενης νομοθεσίας αλλά και ενσωμάτωση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. ενίσχυση δυνάμει του άρθρο 17.1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως όσον αφορά την κοινή ανακοίνωση και την ε, παρέμβαση και συμβολή των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη διαδικασία αυτή της ε, ποιότητας της ε, καταρτιζόμενης νομοθεσίας. Επίσης το πρόγραμμα ε, του ετήσιου και του πολιετούς προγραμματισμού. Επίσης η αρχή της αναλογικότητας, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με βάση και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια σαφή ένδειξη της χρησιμότητας κάθε πρότασης σε όρους ρεαλιστικούς. Στη συνέχεια διαφάνεια και πολιτική υπευθυνότητα σε σχέση με τις απαντήσεις στην ανταπόκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε αιτήματα δυνάμει του 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης μια αξιολόγηση συνολική και κυρίως της ευρωπαϊκής Προστέμενης αξίας, ε, συστηματική και υποχρεωτική ενδεχομένως συμμετοχή των μικρομεσαίων του υπολογισμού της δυνατότητας ανταγωνιστικής ε, και του ωφέλου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, προτάσεις που θα κατατίθενται. Επίσης, διορισμό σε κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές και εκτελεστικές πράξεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στην προπαρασκευαστική εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάγκη για μια διαρθρωμένη ροή ενημέρωσης και πληροφοριών από το Συμβούλιο κυρίως στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Εντοπισμός του ε, gold plating, της αναπομπής δηλαδή πράξεων Επίσης, έλεγχος της στήρησης των διεθνών συμφωνιών και της συμφωνίας τους με, την, με τις συνθήκες, ε, με βάση την ε, νομολογία του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι αν πρόκειται να αλλάξει η νομική βάση μιας Διεθνής συμφωνίας, πρέπει να γίνει συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η επαναδιατύπωση ως νομοτεχνική διαδικασία με στόχο την, τον απόλυτο σεβασμό των ε, όρων των συνθήκων. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την νομοπαραγωγική επιβάρυνση, με αξιόπιστες βεβαίως μεθόδους συλλογή δεδομένων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να αξιολογούν τις ανάγκες και να διαφοροποιούν μεταξύ των ε, του φόρτου που μπορεί με μονομένες προτάσεις να επιφέρουν ε, στα κράτη-μέλη και εν τέλει ο ρόλος των, σωμάτων, ε, των σωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων με βάση τη οργανική μέθοδο. Επίσης, ε, αυτά λοιπόν, περιμένω να βεβαίως να ακούσω τις δικές σας απόψεις Και παρακαλώ την κυρία Ντελβό να προχωρήσει στην ανάγνωση της, ε, του μηνύματος του κύριου Κορμπέτ. Ε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα, συγγνώμη εκ του κύριου Κορμπέτ που δεν μπόρεσε να προσέλθει στη σημερινή συνεδρίαση. Στη συνέχεια να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αλλά και την ε, γραμματεία για αυτό το έργο όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία του νομοθετικού έργου. Το 2016 κάνω μια σειρά συνεδριάσεων μέχρι και από τότε αρχίσαμε και φτάσαμε φέτος και έχουμε διάφορα σημεία τα οποία αφορούν το τι θα καλύψει κάποια έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλίας και θα πρέπει να σας παραπέμψω στο ψήφισμα για ε, το, το ψήφισμα για αυτή τη συμφωνία την διοργανική και θα πρέπει να καταλήξουμε κάπως να βρω την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και έχουμε επίσης κάποια κριτήρια για οριοθέτηση μεταξύ εφαρμοστικών και κατεξοδότηση πράξεων. Ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία και έχει εμπλακεί το Κοινοβούλιο σε κάποιες ε, συζητήσεις για αυτές τις ε, διεθνείς συμφωνίες και επίση είχαμε την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ετήσιο φόρτο. Οπότε σε αυτή την έκθεση υπάρχει μια καταγραφή του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και υπάρχει ενθάρρυνση για τις συνεχιζόμενε διαπραγματεύσει και για την περαιτέρω ε, εφαρμογή τη Διοργανικής Συμφωνία και θα πρέπει να δούμε που επιδέχεται η κατάσταση βελτιώτηση. Και με αυτή την έκθεση δεν θέλουμε να ξανά ανοίξουμε ε, το κουτί της Πανδώρας, δηλαδή να θέσουμε ένα αμφιβόλο την συμφωνία που έχει συναυθεί. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καρίμ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλά. Ε, Μα τα είπε εκ μέρου του Ρίτσαρτ, αλλά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, τότε που θα κάνουμε άλλη μια κοινή συνεδρίαση. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα-δύο πραγματάκια. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πάλι κοινή συνάντηση των Επιτροπών και ανέκαθεν εγώ ήμουν ένθερμος οπαδός του να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κατόφλι να κατέβει κάπως όσον αφορά τις μελέτες των επιπτώσεων και έτσι να υπάρχει περισσότερη προσβασιμότητα για κάποιους πόρους που υποχρησιμοποιούνται. αυτό είναι ένα πολύ εργαλείο, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε περισσότερο. Επίσης, είμαι υπέρ βέβαια αυτών των ε, αξιολογήσεων για τις ε, τροπολογίες και θα πρέπει οι συνεισηγητές να το λάβουν αυτό υπόψη. Επίσης ε, είναι θετικό ότι κάποιοι βουλευτές διστάζουν όσον αφορά αυτές τις μελέτες επιπτώσεων για τις ε, τροπολογίες. Μας φθονούν για τις ωραίες μας τροπολογίες. Να δούμε τι, τι, τι θα μας ωφελήσει τώρα. Να δούμε πώς θα μπορέσει να, να η διαπραγματευτική μας θέση και Όσον αφορά το Συμβούλιο, δεν έχει κάνει καμία αξιολόγηση από ό,τι γνωρίζω. Τίποτα έχουν καθυστερήσει πολύ όσον αφορά την υπόθεση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Οπότε, στις διαπραγματεύσεις να χρησιμοποιήσουμε τις αξιολογήσεις μας, ούτως ώστε να έχουμε ισχυρότερη θέση. φοβούνται τις αξιολογήσεις. Πάντως, οι αξιολογήσεις εκ των υστέρων ωφελούν γιατί έτσι αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα και επιλύονται. Τα είπα και την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τέτοιες ε, αξιολογήσεις αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει και έτσι να ξέρουμε ποια είναι η τελική θέση και τι επιπτώσεις υπάρχουν. Έχουμε τη σχετική μονάδα του Κοινοβουλίου στην προεπικουρικότητα και αναλογικότητα και έτσι μπορούμε να αναλύσουμε σε ποιο βαθμό οι προτάσεις και οι τροπολογίες ε, ε, τηρούν αυτές τις ε, αρχές και αυτό επίσης μπορεί να συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις παρακάτω στάδιο ούτω ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε την συμμόρφωση με αυτές τις αρχές. Και η ανταγωνιστικότητα επίσης είναι κάτι που το έχει μελετήσει η σχετική μονάδα του Κοινοβουλίου ούτως ώστε να αναθεωρηθεί το σχετικό εγκόλπιο που κυκλοφορεί και επίσης θα κάνει και την ερευνά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μείωση του βάρους του φορτίου και εμείς επίσης θα πρέπει να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιοι είναι οι στόχοι και εν τέλει να σας πω ότι συμφωνώ με την ιδέα του να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια για τι εφαρμοστικέ και τις κατεξοδότηση πράξεις και επίση να υπάρχει ε, πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Και σα ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Καρύμ. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να προσθέσει κάτι για το σημείο αυτό. Δεν βλέπω να ζητά κανείς τον λόγο. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της ΑΦΚΟ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Και επειδή η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 9.45, ας κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα λέμε στις 9.45.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 Σα <laughs> ευχαριστώ. So, dear colleagues, can we begin and proceed to the vote? Συνεχίζουμε, λέω πρώτα. Yeah, yes, yes. Συνεχίζουμε και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Πρώτα-πρώτα όμως να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, που είναι το πρώτο σημείο. Let me inform you that today's... Και σας ενημερώνω ότι η σημερινή συνάντηση των συντονιστών ματιώθηκε. Το δε θέμα υπαρθμών 8 πρόκειται να συζητηθεί μετά το σημείο υπαρθμών 4. Υπάρχει κάποια ένσταση, κάποια πρόταση, όχι, επομένως εγκρίνεται η μερισσή διάταξη. 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Σας ενημερώνω. Συμφώνησαν οι συντονιστές για τα θέματα αστικού δικαίου να συζητηθούν στα πλαίσια του διαλόγου των εμπλεκομένων στις 15 ε, Σεπτεμβρίου έχουμε αυτή τη δημόσια διαβούλευση για το διοικητικό δίκαιο και παρακαλούνται όλοι να ενημερώσουν τους φορείς της κοινωνίας, τους ε, πολίτες, τους άλλους εμπλεκομένους. Η δε γραμματεία είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε πληροφόρηση χρειάζεται και πρόκειται τη μέρα που θα αρχίσει αυτή η διαβούλευση να σταλεί ένα email και εκεί θα σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες θα είναι ε, ενημερωμένες. Του παριθμών τρία ήδη το συζητήσαμε, ήταν η κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την ΑΦΚΟ στη 9. Και τώρα συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 4 που είναι η, ψηφοφορία. Έκθεση Άντουσον. Θα γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. One more? Okay. Okay. Yes. Well, anyway, it has been clearly adopted. Είναι σαφής η έγκριση του κειμένου 14-0. Did you vote for or against? Τι είπατε, εκτός μικροφώνου είπε κάτι ο κύριος. Ψήφισατε υπέρ κατά του λέει ο πρόεδρος. Αλλά πάντα εκτός μικροφώνου. Άρα είναι, ψήφισατε υπέρ, άρα είναι 15-0. <laughs> Του Σπάρτακ Ακόμα περισσότερα γκολ από όσο χτες το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Σπάρτακ. Και τώρα έχουμε την έκθεση Χάουταλα. Πάλι ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Όχι. Τι είπατε. Sorry, sorry, Αχ, συμπαθάτε με λέει ο πρόεδρος. Αυτό είναι θέμα προσζήτηση το απόγευμα. Οπότε τώρα ολοκληρώνουμε τις ψηφοφορίες ε, του πρωινού. Okay, okay. So, Λοιπόν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συνεχίσουμε με το σημείο 8. Εξέταση του εγγράφου εργασίας για την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αστικής ευθύνης. Το λόγο έχει η κυρία Μπερζερό, που είναι και η συγγητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν εμφανίστηκε τελευταία. Ξεκίνησε πειραματικά από τις αρχές της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπτύχθηκε στο βιομηχανικό κόσμο από τη δεκαετία του 80. Είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές που ε, βάσει ε, ενός ψηφιακού αρχείου και ενός τρισδιάστατου εκτύπωτη δημιουργεί αντικείμενα. Στην αρχή είχε σχεδιαστεί για να φτιάχνει μοντέλα, πρωτότυπα. Ε, σήμερα αυτά τα μοντέλα αποτελούν τα τρία τέταρτα της αγοράς, της της αγοράς. Χρησιμοποιούνται σήμερα ως υλικά το πλαστικό, ρετίνη και μέταλλα αλουμίνιο χάλιβας, αλλά ήδη βλέπουμε να εμφανίζονται αντικείμενα από ε, ασήμι. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι δυνατή η κατασκευή ε, κοσμημάτων. Όπως σας είπα αρχικά χρησιμοποιητό για την δημιουργία μοντέλων η δυσκολία είναι η, η ταυτόχρονη χρήση πολλών υλικών ώστε να δημιουργούνται τελικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα ας πούμε που είναι το, μισά από πλαστικά, μισά από μέταλλο. Σας έφερα εδώ κάποια αντικείμενα ε, εκτυπωμένα με τρισδιάστατο τρόπο. Εδώ βλέπετε με τεράστια ακρίβεια χιλιοστού, του χιλιοστού ε, βγαίνει το προϊόν έτοιμο, δεν έχει κανείς, κανένα λόγο να το καθαρίσει, να το φτιάξει, είναι έτοιμο για προσπόληση. Χαίρομαι που έζησα μέχρι εδώ για να το δω αυτό. Ε, γίνεται πλέον προσβάσιμη στο ευρύ κοινό αυτή η τεχνολογία με την εισαγωγή των τρισδιάστατων εκτυπωτών που πολλούνται στη Λιανική. Ε, οι υπηρεσίες ε, εξαποστάσεως εκτύπωσης μέσω αρχείων online δίνουν τη δυνατότητα σε όλους για τρισδιάστατη εκτύπωση σε υψηλότερη ποιότητα από ό,τι με μηχανήματα χαμηλού επίπεδου. Η διάδοση των τριζάστατων εκτυπωτών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε συνεργατικούς χώρους εργασίας σε Fab Lab, έτσι όπως το ονομάζουμε αυτό, κατασκευάστηκε σε Fab Lab, ευνοεί την πρόσβαση σε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες τεχνολογίες εχμής χρησιμοποιούν αυτή τη τεχνολογία, διότι βοηθά και την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος. 100.000 ε, αντικείμενα σαν αυτό εδώ, αντί να κατασκευαστούν με ένα τεράστιο μηχάνημα, μπορούν να τυπωθούν με ελάχιστο κόστος, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, με ελάχιστο προσωπικό. Βάζει κανείς απλά τα υλικά στον εκτυπωτή και γίνεται δουλειά μόνη της. Έχει τεράστιες εφαρμογές ε, δυνατές ε, στον ιατρικό τομέα με τη δυνατότητα εκτύπωσης ε, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, ε, ζητάει ο πρόεδρος. Μου είναι αδύνατον, λέει ο μιλήτριο. Ε, είναι δυνατή λοιπόν η κατασκευή οργάνων, ε, μελών του σώματος, Ε, μιλάμε τώρα για μια κατασκευή ε, νεφρού που θα γίνει από ανθρώπινο υλικό για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ε, ως σε κάποιον άνθρωπο ε, και φυσικά και διευθύνται διάφορα θέματα ηθικά για τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων. Ο τομέας της αεροναυπηγικής έχει μεγάλη ζήτηση με τα συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων ε, είναι καταπληκτικό αυτό. Η Airbus έχει ένα αεροσκάφο σε πειραματική φάση αυτή τη στιγμή. Χίλια εξαρτήματά του τυπώνονται διάστατα αυτή τη στιγμή. Η βιομηχανία των ανταλλακτικών επίσης ε, αυτοκινήτων και η βιομηχανία παιχνιδιών αλλά και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών θα επηρεαστούν από αυτή την τεχνική. Δηλαδή, αν σπάσετε ένα εξάρτημα πλαστικό για παράδειγμα στην κουζίνα σας ε, ή σε οποιοδήποτε άλλη οικιακή συσκευή πάτε, στην, ε, ε, πάτε και αντί να παραγγείλετε το εξάρτημα από τον κατασκευαστή πάτε σε κάποιον που έχει ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή και σας το παρέχει εντός 24 ώρου. Η τρισδιάστατη διεκτύπωση και οι σαρωτέ ε, τρισδιάστατη τεχνολογία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ανασύνθεση κατεστραμμένων εξαρτημάτων ή για την ε, ανακατασκευή ε, κομματιών που έχουν χαθεί αρχαιολογικών. Είναι δυνατό δηλαδή να αποκαταστήσουμε για παράδειγμα τους βούδες που κατέστρεψε ο Ντάες και τα λοιπά. Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα και προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα λόγω της, της διάστατης τεχνολογίας ε, ε, συγκεκριμένα ζητήματα ε, νομικά, ασφαλείας, ηθικά και υγείας στον ιατρικό τομέα. Πολλά ζητήματα αφορούν την κατασκευή οργάνων. Εκεί τίθενται θέματα ηθικής όπως της ισότητας πρόσβασης στην υγεία. Τα ζητήματα ασφαλεία είναι πολύ σημαντικά, ειδικότερα όταν μιλάμε για την παραγωγή ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, για ηλεκτρικέ οικέ συσκευέ, για αεροσκάφη και υπάρχει ένα τομέα που εξακολουθεί να μα δημιουργεί ε, ερωτηματικά, είναι τα πυροβόλα όπλα. Κατά την άποψή μου δεν πρόκειται ποτέ να κατασκευάσουμε πυροβόλα όπλα με τρισδιάστατη τεχνολογία. Είναι επιστημονική φαντασία, αλλά είναι κάτι που δεν είναι ε, δυνατό αυτή τη στιγμή. Επίσης μπορεί να διευκολύνει τις ε, δραστηριότητες παραποίησης, κάτι που δυσκολεύει το πρόβλημα, όχι μόνο διότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί σε ιδιώτες εξαίρεση για ε, να φτιάξουν ιδιωτικά αντίγραφα, αλλά διότι μπορεί να διέξαρσει η αγορά ε, παραποιημένων προϊόντων. Για την πρόληψη αυτού λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθεί ε, ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο ώστε το άτομο που παράγει το έργο να μην παραβιάζει τον νόμο και να διασφαλίζει τη σωστή ανταμοιβή του ε, δημιουργού. Η τριζάθετη εκτύπωση όπως καταλαβαίνετε είναι τεράστιας ακρίβειας σε χιλιοστά του χιλιοστού. Δηλαδή αν έχετε ένα ε, γνήσιο έργο τέχνης αντίστοιχης αξίας μπορεί να αντιγραφεί μαζί με την υπογραφή χωρίς κανείς να μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ του γνήσιου έργου και του αντιγράφου. Και αυτό αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα. Εγώ είμαι ευαίσθητη λόγω της δικής μου, του δικού μου επαγγελματικού παρελθόντος, αλλά δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πόσο θα επηρεάσει αυτό τα πράγματα, όχι μόνο στα δικαιώματα δημιουργού, αλλά και στα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αγόρασε ε, ένα γνήσιο εργοτέχνης ε, από κάποιο γνωστό ε, καλλιτέχνη, κάποιο γνωστό γλύπτο από τον Ροντάν, για παράδειγμα, ε, θα μπορεί κανείς να τυπώσει τρισδιάστατα ένα ακριβές αντίτυπο του Ροντάν. Και άνθρωποι που έχουν αγοράσει κομμάτια που κόστησαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, να βρεθούν ξαφνικά με ένα αντικείμενο το οποίο να μην έχει καμία αξία. του Ροντάν ή του Ντρούο λοιπόν. Ε, αυτά περνώ στη συνέχεια. Επίσης τίθενται νομικά ζητήματα που αφορούν και την Επιτροπή μας, ε, ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τη δυνατότητα εξατομίκευσης, ε, προσαρμογής ενός αντικειμένου και εκεί δίνεται θέματα αστικής ευθύνης όσον αφορά τη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο, ακόμη και αν έχει καταθέσει κανείς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ε, αν του προσθέσουμε οτιδήποτε δεν καλύπτεται πλέον από το δικαίωμα διακτησίας. Όσον αφορά την διανοητική ιδιοκτησία πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της εκτύπωση κατοίκων προ ιδιωτική χρήση και την εμπορική εκτύπωση. Ε, καθώς επίσης πρέπει να κάνουμε επίσης και διάκριση ε, της παραγωγής για επαγγελματικού ή για ιδιωτικού σκοπού. Η για ιδιωτικου σκοπου εκτύπωση καθιστά άπειρε, δυνατές άπειρες τροποποιήσεις ε, και προσαρμογές. Αυτές οι νέες τεχνολογίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές ε, στην λειτουργία της αλυσίδα παραγωγής, διότι αρχεία που υπάρχουν ήδη ε, online και η συμμετοχική καινοτομία και τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα μπορούν να βοηθήσουν σε άπειρες και ελεύθερες εξατομικεύσεις και προσαρμογές. Αν πάτε σε ε, ιστοσελίδες με αρχεία ανοιχτού κώδικα, open source, θα δείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ε, καθημερινά χωρίς να το αντιλαμβάνεται καν, πιστεύω, ο δημιουργός του αρχείου. Ε, έχουμε δύο προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις με τους σκιώδες και τους εκπροσώπους της Επιτροπής DG Home Connect και Justice. Εκεί προέκυψε ότι υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά. Αναμφίβολα Σήμερα υπάρχει ένα οπλοστάσιο νομικών κειμένων που μπορεί να καλύψει τα ζητήματα ε, δικαιωμάτων δημιουργού και αστικής ευθύνης και διανοητικής ιδιοκτησίας ε, η νομοθεσία του 2004 για τη διανοητική ιδιοκτησία, για την παραπίση του 2014, για τα υλοτηματικά προϊόντα του 1985. Όλα αυτά τα διαφορετικά ευρωπαϊκά κείμενα μπορούν να καλύψουν ε, την τρισδιάστατη εκτύπωση νομικά. Εγώ συναντήθηκα με πολλούς φορείς ε, της βιομηχανίας, ε, της αγοράς, της τρισδιάστατης εκτύπωσης για να καταλάβω τις τεχνικές και να ενημερωθώ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι επαγγελματίες. Σας, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Σας έφερα κάποια παραδείγματα. Αυτό το ελαττήριο προέρχεται από το κατάστημα Ενό ε, υποδηματοποιού ο οποίο το χρησιμοποιούσε για την ε, επισκευή για, για παπούτσια ε, τώρα παράγει λατήρια για στρώματα τα οποία κοστίζουν 0,10 ευρώ το τεμάχιο και τα παρήγαγε για μια κυρία που έσπασε την πόρτα του ντους πήγε στον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής τη είπε θέλετε 400 ευρώ για ένα τόσο κομματάκι και αυτή πήγε και βρήκε αυτόν τον κύριο ο οποίο τη είπε θα σα κοστίσει ένα ευρώ. Έμεινε πολύ ευχαριστημένη λοιπόν η κυρία αυτή. Ε, δεν είχε καμία διαφορά η αντίσταση του ελαττηρίου ε, ε, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε ατύχημα ε, λόγω ανεπάρξη του ελαττηρίου αναρωτιέται κανείς ποιος είναι υπεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος που σκάναρε το εξάρτημα και το ε, παρήγαγε ξανά στην τρισδέα στο εκτυπωτή του και η κυρία που υπέγραψε ένα συμβόλαιο λέγοντας ότι ο κύριος αυτός δεν έχει κανένα, καμία ευθύνη. Αν τη πέσει λοιπόν η πόρτα στο κεφάλι, ποιο θα φταίει τελικά, δεν ξέρουμε. Στο γαλλικό δίκαιο, όπω δούμε και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκαια, δεν Κανονικά δεν μπορεί κανείς να παραιτηθεί από τις ασκήσεις οποιοδήποτε δικαιώματός του εκ των προτέρων. Ε, οπότε τίθενται κάποια νομικά ζητήματα εδώ, στην πρακτική. Τίθενται. Εγώ με την ευκαιρία του ταξιδιού που κάναμε στο Σαν Φρανσίσκο πήγα να δω το παράρτημα ενός, μιας γαλλικής εταιρείας που ονομάζεται Σκλητεά και, και που παράγει μικρά τεμάχια όπως καρφίτσες, διακοσμητικά, βάζα, πολύ όμορφα. Η, τεχνική, τεχνολογία επιτρέπει να παράγει κανείς καταπληκτικά αντικείμενα. Αυτοί λοιπόν ε, προσανατολιστήκαν ε, στην παραγωγή ανταλλακτικών για drones. Δεν τίποτα, μικρά κομματάκια, ε, ούτε καν ξέρω που μπαίνουν στα drones, αλλά όπως σας έλεγα προηγουμένως, ο, κατα... ο κατασκευαστής ενός ντρόουν χρειάζεται χίλια τεμάχια, όχι εκατό χιλιάδες τεμάχια. Ε, αυτοί λοιπόν παράγουν κάθε μήνα τα χίλια τεμάχια και αυτό κρατά ζωντανές δύο επιχειρήσεις. Δεν είναι και άσχημα. Γίνονται και πολλά άλλα ε, σε αυτή την εταιρεία τη γαλλική που λέγεται Σκελτέ. Βρίσκεται στο Βιλζουίφ και είναι ιδιαίτερα καινοτόμος στο ζήτημα αυτό. Εγώ ρώτησα λοιπόν αυτούς τους επιχειρηματίες ε, για το κατά πόσο αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή νομικά προβλήματα μεταξύ τους και μου είπαν όχι διότι ε, δουλεύουν μεταξύ επαγγελματιών. Κατανέμουν δηλαδή τι ευθύνε τους μεταξύ επαγγελματιών και είναι όλοι τους ασφαλείς. Ε, τώρα τα ζητήματα ασφάλειας και ευθύνης θα δημιουργηθούν όταν θα πουληθούν αυτά τα αντικείμενα απευθείας στα κράτη ή σε ιδιώτες. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι ξεκινάει τώρα μια νέα βιομηχανική εποχή. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι σε 20 χρόνια οι βιομηχανίες, δεν, τα εργοστάσια δεν θα έχουν τη μορφή που ε, γνωρίζουμε σήμερα θα υπάρχουν τεράστια υπόστεγα με τρισδιάστατους εκτυπωτές τεράστιους και όλα θα παράγονται τρισδιάστατα με τρισδιάστατη εκτύπωση. Και αυτό θέτει διάφορα προβλήματα αστικής ευθύνης ε, σε περίπτωση ελαττώματος παραγωγής όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που εμφανίζονται ε, επιλύονται κατά περίπτωση και με συνεννόηση μεταξύ επαγγελματιών. Ο καθένας από αυτούς παρετείται τις ευθύνες του σε περίπτωση παραγωγής αλατοματικού αντικειμένου. Όλε οι νομοθεσίε που έχουμε οριζόντια και εγκάρσια ε, εφαρμογή δεν θα έχουν καμία εφαρμογή στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Πιστεύω λοιπόν ότι από σήμερα θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε να δεν πρέπει να περιμένουμε να, δούμε, να σκεφτούμε ήδη για το τι θα γίνει στο μέλλον, όπως κάνουμε και για τα ρομπότ. Ε, στον ίδιο τομέα βρισκόμαστε ουσιαστικά ε, νομική σκέψη. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα κείμενα τα οποία έχουμε δεδομένων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ε, και καινοτομιών. Εγώ σας έφερα και κάτι άλλο. Μ' αρέσει να δείχνω πράγματα και εδώ θα δείτε τώρα κάτι καταπληκτικό που παρήχθη από κάποιον ε, στους καταπληκτικούς επιστήμονες ε, στο Πανεπιστήμιο της Νάντης. Εκεί υπάρχει ο κύριος ε, Φουρέ, ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε εργατικές κατοικίες και ο οποίος εξελίχθηκε καταπληκτικά από τεχνικός, έγινε μηχανικός και ενδιαφέρθηκε στη, για, τις κοινωνικ... για, το, κοινωνικές κατοικίες ουσιαστικά και σκέφτηκε την κατασκευή λοιπόν μέσω εκτύπωσης τρισδιάστατης. Ε, έχει χτιστεί μια τέτοια κατοικία στην Άντη η οποία θα εγκαινιαστεί τον Μάρτιο. Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χτίστηκε χωρί να υποφέρουν άνθρωποι. Δεν χρειάστηκαν σκαλοσιέ, δεν χρειάστηκε να μεταφέρει κανεί ούτε κουβάδε, ούτε τσιμέντα, ούτε να καταστρέψει την πλάτη του. Ε, εκτυπώθηκε σε... Ε, με τρισδιάστατη εκτύπωση. Έχετε δύο πλαίσια λοιπόν ε, τέτοια και ανάμεσά τους μπαίνει το μπετόν. Και αφού κατασκευαστούν οι τείχοι, μετά αφαίρονται τα πλαστικά υλικά, ε, τοποθείται η μόνωση και δεν έχουν παρά να βάψουν. Είναι καταπληκτική η τεχνική αυτή, από άψη καλλιτεχνική και ε, κατασκευαστική. Χτίστηκε αυτό το σπίτι ανάμεσα σε δέντρα Δηλαδή, αντί να καταστρέψουν δέντρα, έχτισαν το σπίτι ανάμεσα στα δέντρα, χρησιμοποιώντα ε, ένα τριζιάστατο εκτυπωτή. Είναι καταπληκτικό το σπίτι αυτό. Και εγώ του ρώτησα, μα δεν θα χαθούν ένα σωρό θέσει εργασία με αυτόν τον τρόπο. Και μου είπαν, όχι, διότι δεν θα πάψουν ποτέ να χρειάζονται παραθυρα... ε, παραθυράδε, ηλεκτρολόγοι, ε, δουλειέ ωστόσο που δεν δημιουργούν τόση σωματική βλάβη στου ανθρώπου όσο ε, το αυτοί που παθαίνουν οι η Κομισιόν καθυστερεί λίγο, κολυσιεργεί ε, αναμένοντας ε, να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις, να δει τι γίνεται στον τομέα της τρισδιάστατης της εκτύπωσης. Εγώ δεν εκπλήσω. Με πάνω από 5 εκατομμύρια ευαίσθητοι άνθρωποι υπάρχουν ε, σε δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη και η Κομισιόν είπε «Α, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό». Τώρα το διακύβευμα σήμερα τη τρισδιάστατης τη εκτύπωση δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο ρόλος του πολιτικού που θέλει να νομοθετεί είναι να προβλέπει. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των ρομπότ όπως και των τρισδιάστατων εκτυπωτών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελβό έχει στο λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο για την εξαίρετη έκθεση, αλλά και την τόσο ζωντανή και εύγλωτη παρουσίαση. Βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον και προσήλωση τρέφει για τις διάστατες εκτυπώσεις. Βεβαίως, βλέπουμε τις εξελίξεις, τα ρομπότ. Η καινοτομία μας φέρνει ενώπιον νέων προκλήσεων. Βλέπουμε λοιπόν που έχει φτάσει η έρευνα, η πρόοδος, όλες οι προοπτικές, ποιες είναι. Σημεριζόμαστε όσα είπε η Ζωέλα, εγώ προσωπικός. Ασφάλως θα προκύψουν θέματα δεοντολογίας, ασφάλειας. και χωρίς να είμαι τόσο αισιόδοξη για την παρασκευή πυροβόλων όπλων, γιατί αν μπορεί κανείς να εκτυπώσει τρισδιάστατα ανθρώπινα όργανα, γιατί όχι και πυροβολά όπλα. Και άρα η κοινωνία μας βρίσκεται ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Λιγότερο αισιόδοξη μας προς την εξοικονόμηση ενέργειας επίσης. Όλοι οι υπολογιστές και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε καταναλώνουν τεράστια, τεράστιες ποσότητες ενέργειας και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε επαρκείς ενεργειακές πηγές για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Πιστεύω πράγματι ότι θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε στα θέματα της ε, διανοητικής διοκτησίας που είναι της δικής μας αρμοδιότητας αλλά και της δεοντολογίας θα υπενθυμίσω ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας συγκαταλέγεται και η δεοντολογία των νέων τεχνολογιών. Άρα έχουμε να κάνουμε θέματα που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Κατά τρόπο συνεχή. Διανοητική ιδιοκτησία λοιπόν, η πνευματική ιδιοκτησία. Συμφωνώ ότι χρειάζεται να γίνει διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και εμπορικής χρήσης. το καθεστώς ε, στο, το οποίο θα δώσουμε στις πλατφόρμες ανταλλαγών ε, τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Οι προτάσεις είναι καλές. Βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της ε, κατάλληλης αποζημίωσης ή αμοιβή του δημιουργού. Γιατί τρισδιάστατη για το θέμα τη ευθύνη, γιατί να μα απασχολεί σε αυτό, άπαξ και υπάρχει αλυσίδα παραγωγή, ισχύουν οι υφιστάμενες αρχέ στην αλυσίδα παραγωγή, Αλλά ομολογώ πώ δεν με είχε προβληματίσει το ζήτημα των ανταλλακτικών ή άλλων ε, στοιχείων που ενσωματώνονται στο προϊόν κατά τη διάρκεια της επισκευής και που ενδεχομένω αν είναι λατωματικά μπορεί να προξενήσουν ε, ζημία ή σωματική βλάβη στους ε, χρήστες, επιπλέον δηλαδή του έτοιμου προϊόντος. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε τα θύματα, γιατί αυτή είναι η πρωτοαρχική μας ευθύνη και το μέλημα. Σε αυτό λοιπόν πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε. Παρακαλώ τη Ζωέλη να συνεχίσει με το χάρισμα που τη διακρίνει και την αιμονή και υπομονή της και επιμονή της σε αυτή τη δουλειά και πολύ ευχαριστώ και εγώ να την βοηθήσω. Ο κύριος Άξελ Φως. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δύο είναι οι παρεμβάσεις που έχω να σας παρουσιάσω. Η μία είναι εκ μέρους του κυρίου Λούς του Σκιώδου Σιγητού και η άλλη είναι η δική μου. Και μια και έχω αρχίσει στα γερμανικά, σας δώσω τις δικές μου θέσεις πρώτα. Ευχαριστώ καταρχάς θερμά τη συνάδελφο για την ε, πρόταση και την τοποθέτηση είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τη δυνατότητα να, ε, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ύστερα από μια τόσο ζωντανή παρουσίαση. Συνήθως ε, έρχεται με βραδιπορία η ε, αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων και των εξελιξιών τους από τον νομοθέτη. ωστόσο, συμφωνούμε με τα όσα είπατε εν γέννη, είναι καλές οι προτάσεις. Στα όσα επεσήμανε η κυρία Ντελβό ήδη, επί παραδείγματι την τρισδιάστατη εκτύπωση πυροβόλων όπλων ή, ή οδήποτε άλλου όπλου, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συμπληρώσουμε το εξή ότι θα μπορούσαμε να ε, εκτυπώσουμε ακόμα και τρόφιμα κατά τρόπο τρισδιάστατο το ε, ψηφιακό ή το τρισδιάστατο μπέργκερ έχει ήδη ε, εκτυπωθεί, οπότε έχουμε άλλα ζητήματα. Για δε την εγκληματικότητα, εδώ ε, έχουμε πολλά ζητήματα και μάλιστα αναφέρομαι όχι μόνο στα ανταλλακτικά γιατί στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν έλεγχο της κυκλοφορίας των όπλων ε, από το κράτος ενώ τώρα αν υπάρχει δυνατότητα της τρισδιάστατης εκτύπωσης ο γείτονα μου να αποφασίζει ότι χρειάζεται όλο και περισσότερα όπλα, τα οποία μπορεί να εκτυπώσει τον τριζάστα του ε, εκτυπωτή του και μάλιστα αυτά θα λειτουργούν και όλα. Τότε έρχεται μια τελείω διαφορετική ε, ε, διαμόρφωση πραγματικότητα. Έρχεται ένα διαφορετικό κόσμο τελείω μπροστά μα. Το ίδιο και για τα ναρκωτικά, εάν μπορούμε να εκτυπώσουμε τρισδιάστατα ναρκωτικά. Δηλαδή μπορεί κανείς να δημιουργήσει στο σπίτι του, στην αποθήκη του ή στο ε, υπόγειό του ε, πράγματα τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία. Το ίδιο και με την εκτύπωση, εκτύπωση ανθρώπινων οργάνων. Πολύ ωραία αναφέρθηκαν όλα αυτά τα επιχειρήματα, αλλά από την άλλη βιολογικά ή χημικά όπλα, μήπως θα είναι και αυτό δυνατόν να εκτυπωθούν. Και αυτά δυνατόν να εκτυπωθούν. Γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος αυτών των ψηφιακών και μάλιστα και, του, και του, των οδηγών εκτύπωση, το πώ θα γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια εύκολη λύση βεβαίω, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτά τα ηλεκτρονικά ε, έγγραφα να τα ελέγχουμε. Τα πυρηνικά όπλα, παραδείγματι, μέχρι τώρα ανήκουν στον ε, απόλυτο κρατικό έλεγχο. Εάν αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν, ε, όμω θα φτάσουμε και σε αυτά στην τρισδιάστατη εκτύπωση επαναστατική εξέλιξη ασφαλώς. Και βεβαίως θα ήθελα η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο μας να μπορέσει να χαράξει πρωτοπόρο, ε, πρωτοπόρες θέσεις για τα θέματα αυτά της, της διάστατης εκτύπωσης. Ασφαλώς θα πρέπει να μας απασχολήσουν και άλλα θέματα, αλλά όλα αυτά θα χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο οπωσδήποτε. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας αναγνώσω την παρέμβαση του κυρίου Λούις Δεγκράντες στα αγγλικά αυτή τη φορά μια ναι, και με παρακάλεσε να τον ε, εκπροσωπήσω σήμερα. Το έγγραφο εργασίας της Ζωέλ Μπερζουχόν αξίζει θετική αξιολόγηση. Πρόκειται για μια ε, αποτελεσματική διάγνωση των προβλημάτων της τρισδιάστατης εκτυπωτικής διαδικασίας, αλλά βεβαίως χρειάζεται πιο λεπτομερής έκθεση λόγω Τη σημασία που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογία και μάλιστα λόγω όλων των τομέων που αυτή καλύπτει. Ιδιαίτερα η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να γεννήσει ζητήματα υγείας, ασφάλειας αλλά και νομικά πάρα πολύ σημαντικά, όπως και εγκάρσια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διανοητική, πνευματική διοδιοκτησία, την αστική ευθύνη, ε, θέματα δηλαδή που ανήκουν στο πεδίο ε, αρμοδιοτητών της Νομικής Επιτροπής σε σχέση με τη διανοητική ε, ιδιοκτησία ή ο σχεδιασμός πρωτότυπου ε, εγγράφ αντικειμένου και η εκτύπωσή του τρισδιάστατα είναι μια πρώτη προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την κάλυψη των διαμεσολαβητών στην διανοητική ιδιοκτησία. Επίσης, ο περιορισμός της αστικής ευθύνης, ακόμα τουλάχιστον σε, στο βαθμό που κάποιος δεν έχει ενεργό ρόλο στο, στην αποθήκευση των αρχείων και δεν μπορεί να υπάρχει περιορισμός. Χρειάζεται λοιπόν να διευκρινιστεί η νομοθεσία για την αστική ευθύνη συγκεκριμένα και την λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας για να εξετάσει αν αυτή καλύπτει τις υφιστάμενες ανάγκες με βάση και το βαθμό ζημίας που μπορεί να προξενήσει ένα αντικείμενο που έχει παραχθεί με την τρισδιάστατη τεχνολογία και γιατί θα είναι δύσκολο ίσως ο ιδιώτης να εντοπίσει τον παραγωγό κατασκευαστή αυτού του αντικειμένου ή εξαρτήματος. Ο παραγωγός του λογισμικού με βάση το οποίο λειτουργεί, αν θέλετε λίγο πιο γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος, α, συγγνώμη, λίγο πιο αργά. Μάλιστα, τρισδιάστατος εκτυπωτής, τελεία. Για να ολοκληρώσουμε από την κατασκευή-παρασκευή του αντικειμένου οι δυνατότητες σχεδιασμού και εφαρμογής του είναι απεριόριστες. Οι φυσικές, υλικές μάλλον και λοιπές ιδιότητες του μπορούν να επηρεάσουν και τον τρόπο λειτουργίας της αλυσίδας παραγωγής. Η δε τα δε αρχεία ανοιχτή πηγή μπορούν να διαμορφωθούν κατά τρόπον ώστε να τροποποιηθούν και άρα υπάρχει ευρύτερη πρόσβαση του κοινού. Ε, η αντιμετώπιση των παραβιάσεων διανοητική ιδιοκτησία θα πρέπει να καλυφθεί από νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ή προσαρμογή τη υφιστάμενης νομοθεσία συγκεκριμένα για την τρισδιάστατη εκτύπαση, νομοθετική αντιδράση και αντιμετώπιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες και έργα, ε, να υπάρχει επαρκής υποστήριξη και όχι παρεμπόδιση της τεχνολογίας από την νομοθεσία. Thank you well. Ε, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μείνει κατάπληκτος από όλα αυτά τα νέα πράγματα, αυτή την καινοτομία, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη νέα τεχνολογία. Για να δούμε πρώτα πρώτα τι μας είπε ο κύριος Λουίς ε, Γκράντες, ε, όπως τα ακούσαμε από τον συνάδελφο Φως το δίκαιο, ο νόμος δεν είναι δυνατόν να αποτελούν φραγμό στην τεχνολογική ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους μηχανισμού ρυθμιστικού που να ε, περιχαρακώνουν ε, αυτές τις ε, εξελίξεις. Γιατί αλλιώς πρέπει να πω ότι φόβο προκαλούν οι ανακαλύψει ανακαλύψεις, νέε εφευρέ. Πάντως εγώ τρέφω αισιοδοξία για όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι έχει αναφεί κάποιο καινούριο πρόγραμμα που δεν το έχουμε ξαναδεί σε άλλους τομείς της εξέλιξη εξέλιξης ε, εξορισμού το δίκαιο είναι αργό. Ε, αργεί να προσαρμοστεί στις ανακαλύψεις, στις εφευρέσεις ε, και βέβαια είναι ακόμα και πιο εφάνταστη, πιο εφευρετικοί οι εγκληματίε. Και οι νομικοί ακολουθούν ακολουθούν το έγκλημα, αργούν να προσαρμοστούν και αυτό έχει σχέση και στο πεδίο της οικονομίας όσο και στο πεδίο της επιστήμης. Αυτό το λέω γιατί έχουμε εδώ πέρα κάποιες θετικέ πλευρές του θέματος, θέματα που ωφελούν τον πολίτη. Να, να σας πω και εμένα τι μου έχει συμβεί. Χάλασε ένα φανάρι στο αμάξιμο και ε, τι έγινε, έλειπε ένα ανταλλακτικό. ένα, ένα μικρό κομματάκι εξάρτημα που θα στήριζε ε, την, την λάμπα. Τέλο πάντων πήγα και αγόρασα το σετ, αλλά πάντως υπάρχουν κάποιοι κατασκευαστές που καταχρώνται τις θέσεις που έχουν στην αγορά και έδωσα ένα σωρό λεφτά και όλα αυτά έδωσα ξέρω 200 ευρώ ενώ το κομματάκι το οποίο μου έλειπε θα έκανε ένα-δυο ευρώ. Να επομένως Πώ με τη νέα αυτή τεχνολογία μπορούμε να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδου καταχρηστικές συμπεριφορέ. Οπότε έτσι βέβαια λέμε μπορεί να παραχθούν και όπλα ε, σήμερα πάντως. Αγοράζει κανείς ό,τι θέλει στην αγορά. Ό,τι όπλο θέλει μπορεί να το βρει στην αγορά. στην Αμερική ακόμα και στο σούπερ μάρκετ που λένε τα όπλα. Επομένω, αυτό το οποίο τώρα χρειάζεται είναι να υπάρχει κάποιο είδου παιδεία, για τους νέους. Θα πρέπει να έχουν δουλειά, θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές συνθήκε, ούτω ώστε να συμμετέχουν όλοι, να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και να μην στρέφονται στην εγκληματικότητα. Τώρα όσον αφορά τα καλλιτεχνικά έργα Εντάξει, έχουμε κάποια γλυπτά, έναν μπούστο του Ναπολέοντα, ε, του Μπετόβεν. Ναι, φυσικά και πάντοτε θα ισχύει η μεγάλη αξία του πρωτοτύπου. Καλά, θα μπορούσε κανείς σε διάφορα υλικά, σε μάρμαρο, βασάλτη, να φτιάξει τα αντίγραφα. Οπότε, συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να τρέφουμε αισιοδοξία θα πρέπει να υποστηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, να τις προωθήσουμε, να τις εξελίξουμε και ταυτόχρονα όμως να προβλέψουμε και κάποιους ε, ε, μηχανισμούς ώστε να προστατευτεί ο κόσμος από την κατάχρηση, ε, από την κακή χρήση τέτοιων ε, εφευρέσεων. Χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται ενημέρωση και απασχόληση για όλους. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα όπως και συνάδελφοι να ευχαριστήσω θερμά την συνάδελφο Μπερζερών γιατί με ενθουσιασμό, με νεανικό ενθουσιασμό αγκάλιασε αυτό το ε, θέμα. Πολύ ευχαριστώ αυτό να βλέπουμε ένα τέτοιο θετικό πνεύμα που διαπνέει το, την έκθεση και γενικότερα το έργο της. Σύμφωνα με τους αδέλφους και ιδίως με τον ε, ε, Αντώνιο Πίντο ότι δεν έχουμε τώρα κάποιο πρόβλημα που τώρα ανοιχθεί. Τα ξέρουμε αυτά. Ήδη. Ξέρουμε το τι νομική πλαισίωση μπορεί να γίνει για τέτοιες εφευρέσεις. Από τότε που εφευρέθη ο ηλεκτρισμός έχουμε το ζήτημα. Οπότε βλέπουμε επίσης ε, τι προβλήματα έχουν αναφεί με την ε, τεχνητή ευφυΐα, με την ψηφιακή τεχνολογία, οπότε το ίδιο τώρα προκύπτει και με αυτή την τρισδιάστατη εκτύπωση. Οπότε και αντίστοιχα ξέρουμε τι προσέγγιση σόφρονα θα κάνουμε, όπως και με τα ρομπότ. Εκεί είχαμε κάποιες διχογνωμίες, αλλά ούτε αυτό είναι πρόβλημα έτσι και αλλιώς. Υπήρξε σύγκληση απόψεων και στην έκθεση Ντελβό για το κατά πόσον θα υπάρχει νομική προσωπικότητα για τα ρομπότ ή δεν θα υπάρχει και τελικά ποιος φέρει την ευθύνη όταν υπάρξουν κάποια προβλήματα, ατυχήματα, ε, προστριβές, τέλο πάντων κάτι αρνητικό για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι από πλευράς ηθικής. Να δούμε, όπως και στα άλλα δύο θέματα που σας είπα, τη τεχνητή ευφυΐα, ρομπότ και ψηφιακά, ποια είναι τα προβλήματα, τι γίνεται για την πνευματική διευθυνσία. Θα πρέπει οι διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ε, πιστοποίησης, της ε, αυθεντικότητας, οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τον έλεγχο, με την καταπολέμηση της απάτης. Να μιλώ για την υπηρεσία των ε, βρεστεχνιών του Αλικάντη και του Μονάχου, που το παρατηρητήριο λοιπόν που είναι στην Ισπανία, στο Αλικάντη. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν, θα πρέπει να παράξουν το ΣΥΠΗΝ ή να μας δώσουν το, το υλικό που χρειάζεται για την νομοθεσία. Είναι θέμα πραγματική ιδιοκτησία και είναι και το θέμα της ε, ευθύνη. Θα πρέπει επομένω με προσοχή να προχωρήσουμε, αλλά επί τη βάση τη ε, αρχής. Να, να τα ζυγίσουμε όλα. Πραγματική ιδιοκτησία, ευθύνη κλπ. κλπ. Επομένως να φτιάξουμε ένα πρώτο κείμενο που να πλαισιώνει αυτέ τι νέε εφευρέσει και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Επίσης ε, κάτι άλλο πέραν των ηθικών θεμάτων, πέρα από τα θέματα δημοτικής ιδιοκτησίας και ευθύνης. Τέταρτο θέμα. Οι οικονομικές συνέπειες. Να είπαμε για, τα, για τις οικοδομές, είπαμε για αυτά τα μεγάλα αντίγματα που μπορούν τώρα να κατασκευαστούν. Όλα αυτά μας βάζουν σε, μια καινούργια φάση στην οικονομία. Θα έχουμε καταβήθηση των, των τιμών. Οπότε τέλος πάντων ευχαριστώ τη συνάδελφα. Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια, μια πρώτη έκθεση Πρόκειται για κάτι το οποίο πάρα πολύ θετικά ε, ε, χαρά και ενθουσιασμό το προσεγγίσατε. Μπράβο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, όχι, όχι, όχι. Ο κύριο Άντερσον πρώτα θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τρισδιάστατη εκτύπωση ως τεχνολογία περιλαμβάνει τεράστιες δυνατότητες. Πολλά υπόθηκαν, αλλά ως πράσινος πρέπει να επισημάνω ότι μπορεί να δημιουργήσει τεράστια πλέον εκτήματα για το περιβάλλον. Ε, θα εξοικονομηθούν πόροι μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές. Επίσης ε, θα δώσει τη δυνατότητα ε, παραγωγής εξαρτημάτων για την επισκευή προϊόντων θα μπορεί να τα παράγει κανείς μόνος του ή θα μπορεί κανείς να αποταχθεί σε μια μικρή επιχείρηση που θα παράγει εξαρτήματα κάποια για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν μέσω τρισδιάστατης τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραχθεί εκ νέου ένα προϊόν. Αντί να αντικαθιστάμε λοιπόν μπορούμε να επισκευάζουμε. Είναι πολλά υποσχόμενη λοιπόν αυτή η τεχνολογία. Ε, επίσης θα βοηθήσει να μειωθούν τα κόστη μεταφοράς ε, και οι ανθρακούχες εκπομπές λόγω των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Θα παράσχει τεράστιες δυνατότητες σε μεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν ε, στον τομέα των επισκευών. όταν δεν έχουν στο αποθέμα τους όλα τα μικροεξαρτήματα που χρειάζονται. Ε, φυσικά αυτό θα φέρει τεράστια κέρδη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τα θέματα ε, ευθύνης και λογοδοσίας και ηθικής. Αναφέρθηκε η παραγωγή όπλων, πυροβόλων όπλων μέσω τρεις διάστατης εκτύπωσης. Εγώ θα αποθάρρυνα άπαντες από τέτοια παραγωγή μέσω της τρεις ε, τεχνολογίας. Είναι επικίνδυνο αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Ωστόσο είμαι αισιόδοξο ε, όσον αφορά τις ε, τεχνολογικές υποσχέσεις, ε, παρατηρείται βελτίωση της κατάστασης συνήθως και πολύ συχνά γρήγορη βελτίωση. Οπότε Οπότε, ξέρετε, αυτά τα όπλα για τα οποία συζητάμε μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνα, να δίνουν λύσει. Ε, ξέρουμε ούτω ή άλλω ότι τέτοια όπλα υπάρχουν. Ε, το θέμα τη λογοδοσία επίση είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Απαιτείται επίσης και μια προσέγγιση ε, φιλική προς την καινοτομία στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πολλά καλά μπορούν να προκύψουν, οπότε θα, θα πρέπει να προσέξουμε να μην θεσπίσουμε θεσμικούς κανόνες που να περιορίσουν την καινοτομία. Ας δούμε το ζήτημα της διανοητικής ιδιοκτησίας, του copyright. Έχουμε ήδη σχετική νομοθεσία, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε ήδη δυσδιάστατους εκτύπωτες που αρχίζουν να είναι πολύ πολύ αποτελεσματικοί Ε, μπορούν καλλιτέχνες ε, να τυπώσουν έργα τέχνης για παράδειγμα. Είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο όπου κάποιοι καλλιτέχνες βγάζουν περισσότερα χρήματα από τα έργα τέχνης τους πουλώντα δυσδιάστατα αντίτυπα των έργων τους. Η νομοθεσία που έχουμε σήμερα καλύπτει ήδη αυτά τα έργα και θα πρέπει να προσέξουμε να μην εισαγουμε νέου κανόνε ε, που θα περιορίσουν την κοινοτομία. θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν που δεν αναλύονται πλήρω σε αυτή την έκθεση, αλλά τουλάχιστον αναφέρονται. Η πιθανή επιβολή φορολογία στην τρισδιάστατη ε, εκτύπωση ω ως αποζημίωση των κατόχων των αρχικών δικαιωμάτων ε, για προστασία τους από τα παράνομα αντίγραφα. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη επιφύλαξή μου. Έχουμε ήδη ένα σύστημα ε, τελών ε, για αντίτυπα που επιβάλλεται σε ανθρώπους κατόχους υπολογιστών υπολογιστών ή γενικώ μηχανημάτων όπου είναι δυνατή αποθήκευση κάποιων πραγμάτων για παράδειγμα ε, τα κινητά τηλέφωνα είναι πιο ακριβά διότι ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία ισχυρίζονται ότι το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αρχείων μουσικής. Ε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Θα το διορθώσουμε με το χρόνο. Θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην εισαγούμε οποιαδήποτε πρόταση που να αποδειχθεί επιβλαβή για την κοινοτομία. Επίσης αναφέρεται το νομικό όριο στον αριθμό των αντιτύπων ή αναπαραγωγών. Εγώ θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτή την πρόταση, διότι ξέρετε εδώ αυτό μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Όποιο πάει να μου περιορίσει τον αριθμό των βιβλίων που θα έχω στη βιβλιοθήκη μου, εγώ θα φέρω μεγάλη αντίσταση. Τέτοιε προτάσει λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε καλά αυτά που λέει η συγκήτρια και πρέπει να υπάρχουν και κάποια καλά στοιχεία σε όλα, ακόμη και στα, σε αυτά που ανέφερα ω αρνητικά, διότι ναι, προβλήματα θα υπάρξουν όπω αναφέρθηκε. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, ε, τα μηχανήματα τρισδιάστατη εκτύπωση για εγκληματικέ δραστηριότητε και θα πρέπει να έχουμε κάποια δομή που να το εμποδίζει αυτό, Όπω για τα πάντα. Άλλα δύο πραγματάκια που θα ήθελα να πω η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικό εργαλείο παραγωγής ε, έργων τέχνης. Η ελευθερία καινοτομία ε, θα βοηθήσει τους καλλιτέχνες. Δεν πρέπει να ε, τους περιορίσουμε. Και τέλος ήθελα να πω κάτι για τα αρχαία ανοιχτού κώδικα, για τα open source files. Αυτά τα αρχεία στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης αρχίζουν να αποτελούν ένα κοινό αποθετήριο χρήσιμο για όλους. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την ανάπτυξη των καλών βιβλιοθηκών αρχείων open source που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. Θα αποδειχθεί πολύ επωφελής για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε επωφελές στο διαδίκτυο, πολλοί υπολογιστές ήδη τρέχουν με προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Ε, και πιστεύουμε ότι και στον τομέα της διάστασης της θα αποβούν τεράστιο ωφέλους για την κοινωνία. Ευχαριστώ κυρία Ρέντα. Αγαπητοί φίλοι, έχω πολύ καλές ειδήσει. Δεν εξωτερώνει τους κανόνες θερμοδυναμικής ο τρισδιάστατος εκτυπωτής. Μπορεί να εκτυπώσει δηλαδή κανείς μόνο αυτό για το οποίο έχει και τις πρώτες ύλες. Άρα όλα αυτά που σας φοβίζουν, πυρηνικά όπλα, ε, ναρκωτικά και ούτε καθεξής δεν μπορεί κανείς στο σπίτι του να τα εκτυπώσει τόσο εύκολα. Μόνο αν έχει στη διάθεσή του σε σκόνη τα ναρκωτικά μπορεί κανείς να τα μετατρέψει σε χάπι μέσω ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή. Και για τα όπλα το ίδιο ισχύει. Ε, πρέπει να έχει κανείς δηλαδή τις πρώτες σύλλες στη διάθεσή του. Επομένως ο εκτυπωτής τον οποίο μπορεί κανείς να πάρει και να βάλει στο σαλόνι του ε, μόνο με πλαστικό μπορούν να κάνουν εκτύπωση και και όπλα από πλαστικό δεν ε, λειτουργούν. Βεβαίω και μπορεί να υπάρξει τρισδιάστατο εκτυπωτή που κάνει πιο ε, σοβαρή παραγωγή και μπορεί να φτάσει μέχρι το όπλο, αλλά και εκεί χρειάζονται και τα βλήματα, χρειάζεται το μπαρούτι, χρειάζονται οι σφαίρες και αυτά. Η πρώτη ύλη, το μπαρούτι, ε, η πυρίτιδα, είναι αυτό που απαιτείται για να σχηματιστεί μια σφαίρα, ακόμα και με τον καλύτερο τρισδιάστατο εκτύπωτη. Άρα χωρίς πυρίτιδα τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο εκτυπωτής. Άρα κάπου πρέπει να ψάξει κανείς να βρει την πυρίτιδα και αυτό είναι υπό αυστηρό έλεγχο ασφαλώς το ίδιο και για τα πυρηνικά όπλα. Τρισδιάστατη εκτύπωση ε, πυρηνικών όπλων θα σήμαινε ότι ε, θα ήταν επικίνδυνη αν μπορούσα να, βγω στο, να μπω στο Amazon, στο site του Amazon και να αγοράζω πλουτόνιο εμπλουτισμένο. Δεν είναι αυτό όμω. Εδώ μην, μην φαντάζεστε κάτι σαν το Star Trek που επιτρέπει να ε, εμφανιστεί μαγικά ε, ένα προϊόν χωρίς πριν να υπάρχει τίποτε. Όχι, απαιτούνται πρώτες ύλες, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι <clears throat> δεν υπάρχουν ε, τέτοιες ε, δυνατότητες, αλλά μην φανταστεί κανείς ότι μπορεί κανείς να, κάνει, να εκτυπώσει ναρκωτικά τρισδιάστατα χωρίς πρώτη ύλη, να τα βάλει σε ένα φλιτζάνι του τσαγιού και να το σερβίρει σε κάποιον. Δεν έχει φτάσει μέχρι και η τεχνολογία. Η Επιτροπή έχει τίποτα να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ από την DG Just, από την ε, Μονάδα Ενοχικού Δικαίου. Ευχαριστούμε καταρχάς ε, την Επιτροπή σας που ασχολείστε με την τρισδιάστατη εκτύπωση για τη σημαντική δουλειά της μέχρι τώρα, δουλειά για την οποία τρέφουμε βαθύτατη εκτύπωση, ε, εκτίμηση και παρακολουθούμε εκ του σύναγγες. Επίσης, ε, παρακολουθούμε γενικά τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω εξελίξει Η τρισδιάστατη εκτύπωση, ιδιαίτερα υπό το φω της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, οδηγία που θα καλύπτει ορισμένες πτυχές ενοχικού δικαίου και συμβάσεων σχετικών και θα πρέπει να σας πω ότι μια χαρά τα πάμε μέχρι τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ρητά στην τρισδιάστατη εκτύπωση, στην αιτιολογική σκέψη 16 αναφέρεται ότι αυτή η, οδηγία, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται και, στους, ε, και στα files ε, που καλύπτουν και το λογισμικό τρισδιάστατο της εκτύπωσης, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην ρύθμιση της τεχνολογίας ή τη ζημία που προξενείται από την χρήση αυτής. Άρα πρέπει τώρα να διευκρινιστούν τα ζητήματα τα οποία έχουν ε, αφαιθεί εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και άλλα ζητήματα ε, Αντικειμενική ευθύνη που δεν καλύπτονται μέχρι τώρα από την νομοθεσία και γι' αυτό προσβλέπουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ανάλυση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο του θέματος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κλάουδια Μαρτίνεθ Φέλεξ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, από την ε, DG Grow αναπληρώτερα τμήματάρχης του τμήματος που ασχολείται με την οδηγία τη σχετική με την ευθύνη από αντικείμενα, από προϊόντα. Τα αντικειμενική ευθύνη από προϊόντα ελαττωματικά καλύπτει και την τρισδιάστατη εκτύπωση και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εξετάζει με τόση προσοχή την τρισδιάστατη εκτύπωση. Ένα από τα προϊόντα που μας απασχολούν, που εξετάζουμε και στο πλαίσιο μελέτης που πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί και αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της οδηγίας για την αντικειμενική ευθύνη που έχουμε ε, προετοιμάσει. Εξετάζουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μία προσέγγιση για τα προϊόντα αυτά που να δίνει ισορροπημένες απαντήσεις τόσο για τον καταναλωτή καλές όσο και για την καινοτομία ικανοποιητικές. Τα απορίσματα της αξιολόγησης οδηγίας για την αντικειμενική ευθύνη θα κατατεθούν σύντομα μέσα στο 2018, στις αρχές του 2018 συγκεκριμένα. και το Κοινοβούλιο θα ε, τηρηθεί ενημερό. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Οπότε ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το σημείο αυτό. Εκτός αν η κυρία Μπεζερόν θέλει να δευτερολογήσει. Όχι, όχι, δεν έχουν προσθέσει ό,τι λέει η κυρία Μπεζερόν. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. είναι τόσο θετική και συμφωνώ με την ε, ε, με τον συνάδελφο εδώ. Και για τα όπλα έχετε δίκιο, φτιάχνει ο άντρα μου πάρα πολύ εύκολα όπλα, παίρνει ένα σωλήνα κλπ. Όχι, όχι, δεν, δεν θα φτιάξουμε όπλα με τον εκτυπωτή τον τρισδιάστατο και για τα ατομικά όπλα τα είπαμε. Τώρα για τον κύριο Ντεγκράντες, ναι, συμφωνώ, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία, η οποία όμως να μην φρενάρει τις εξελίξεις. Πρόκειται για αξιοσημείωτη πρόοδο. Ε, αυτό εκπροσωπούν ε, αυτοί οι εκτύπωτες. Επίσης, ε, ναι, όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κοιτάξτε το, τελικά είναι περιορισμένη η ζήτηση των ανταλλακτικών ε, γίνονται επί παραγγελία. Οπότε σε σχέση με την μαζική παραγωγή έχουμε εξοικονόμηση ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Συνεχίζουμε τώρα με το σημείο υπαριθμών 5. Παρουσίαση τη μελέτη για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για το καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων. Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ελοντιτήριον από την ε, υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης για την ε, αξιολόγηση αυτών των κοινωνικών αλληλεγγύων επιχειρήσεων. Ζήτησε η Επιτροπή σας από την Υπηρεσία Έρευνας του Κοινοβουλίου να συντάξει αυτή την αξιολόγηση, ούτω ώστε να υποστηρίξουμε την νομοθετική πρόταση για αυτές τις εταιρείε. Και κάναμε στην υπηρεσία μας αυτή την μελέτη, αυτή την αξιολόγηση και για το τι νομοθετική δράση θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Εκεί επισημαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα στο ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και λέμε ότι σε νοσιακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει και μπορεί να υπάρξει προσθεμένη αξία. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να δημιουργήσουμε με συντονισμό τέτοια προσθεμένη αξία. Πρώτα πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι μόνο κάποιοι από τους παίκτες σε αυτόν τον ε, χώρο κοινωνικής οικονομίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, αλλά θα πρέπει πρώτα πρώτα να δούμε το θέμα του ορισμού. Δεν υπάρχει όμως ε, ορισμός ο οποίος διεθνώς να βρίσκει όλους σύμφωνους, όμως εδώ στην Ευρώπη έχουμε συγκλίνει σε έναν ορισμό επί τη βάση εννέα κριτηρίων. Ε, τρεις ομάδες των τριών κριτηρίων, τρεις, τρεις, εννιά, πρώτα-πρώτα, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχή δραστηριότητα για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο οικονομικού κινδύνου και θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό αμοιβωμένη εργασία. Τώρα, όσον αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να είναι ε, ρητά ο εκπεφρασμένο σκοπό τη να ωφελήσει την κοινότητα, την κοινωνία, ε, να είναι μια πρωτοβουλία από ομάδα πολιτών και να υπάρχει ε, διανομή περιορισμένου κέρδους. Να έχει επίσης υψηλό βαθμό αυτονομίας, να μην στηρίζεται η λήψη των αποφάσεων σε κατοχή κεφαλαίου και να υπάρχει συμμετοχή φύση. Οπότε βλέπουμε ότι πρώτα στηρίζονται σε πάρα πολλού τομεί, όπως είναι ε, το να ωφεληθούν οι μη προνομιούχοι και κοινωνικές υπηρεσίες, ε, περιβάλλον, ε, παιδεία, πολιτισμό, τουρισμό και δραστηριότητε αθλητικέ. Οπότε έτσι υπάρχει πραγματική συμβουλή στην οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε όλο ένα και περισσότερε τέτοιε εταιρείε και υπολογίζονται μεταξύ 130.000 και 250.000 τέτοιων κοινωνικών επιχειρήσεων ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δε θεσμικά τη Ένωση έχουν αναγνωρίσει αυτέ τι σημαντικέ επιπτώσει που υπάρχουν για την ανάπτυξη τη Ένωση. Αυτό επανειλημμένα και έχουμε πάνω από 200 ε, έγγραφα τη Ένωση τα οποία έχουν συνταχθεί σε σχέση με αυτό τα τελευταία χρόνια. Και εκεί τονίζεται ότι η συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά παραμένει περιορισμένη. Όντω ε, αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων. Όπω το ότι δεν υπάρχει κοινή κατανόηση ε, του, του, του τι θα πει κοινωνική οικονομία. Δεν προβάλλονται. Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση ε, και σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Μόνο 18 κρατημέλη έχουν συγκεκριμένη νομοθεσία που αναγνωρίζει και ρυθμίζει τα των κοινωνικών επιχειρήσεων και σε κάθε κράτος υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις Έχουμε δύο τέτοιε μορφέ, Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομική μορφή σε σχέση με την νομική δομή μια τέτοια ε, επιχείρηση και σε άλλα κράτη-μέλη προβλέπεται ε, ένα νομικό καθεστώ το οποίο μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένες νομικές μορφές αλλά πρέπει να πληρώνονται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Επομένως, αυτό το πρόβλημα σημαίνει ότι έχουν δυσκολία αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση αλλά και στις αγορές και έτσι δεν μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις δραστηριότητά τους. Θα πρέπει επομένως να δούμε ότι έχουν δυνατότητες να επεκταθούν σε άλλες αγορές. 56% τέτοιων επιχειρήσεων έχουν τέτοιες προσδοκίες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στο Μήνο Βασίλειο, το ποσοστό των εργοδοτών τέτοιων επιχειρήσεων ε, αυξάνει και θα πάει στο 78%. Πάντως, έχουμε όλες αυτές που πρέπει να επεκταθούν τις επιχειρήσεις, αλλά μόνο λίγες το καταφέρνουν. Για παράδειγμα, στη Γερμανία. Μόνο 6% των κοινωνικών επιχειρήσεων λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σκωτία, μόνο 7% των κοινωνικών επιχειρήσεων συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις ε, οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν ε, θεμητές ε, συνθήκες συνταγωνισμού, ισότητα ευκαιριών, να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση της δραστηριότητας τους ακριβώς, να πρέπει να έχουν και κάποια νομικά μέσα για να μπορέσουν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες τους διασυνοριακά. Οπότε το πόσο θα ωφελήσει ένα τέτοιο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το περιεχομένο του. Έχουμε οικονομική προστιμένη αξία. Θα έχουμε οικονομίες κλίμακα για αυτέ τι επιχειρήσει. Μπορεί αυτέ οι επιχειρήσει να ωφεληθούν από πρόσβαση με μεγαλύτερη αγορά και από μεγαλύτερη προβολή του. Επίση θα υπάρξει και αποτέλεσμα μόχλευση στα κράτη-μέλη εκεί που δεν υπάρχει ή είναι πολύ σκιώδε το νομικό πλαίσιο. Και ε, έτσι θα ενθαρρυνθούν αυτές οι επιχείρησεις να καινοτομήσουν και με αυτό το πλαίσιο θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για υπηρεσίες και αγαθά που παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και τέλος, ένα τέτοιο πλαίσιο θα βοηθήσει αυτές τις εταιρείε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, θα τους ενισχύσει τα πλεονεκτήματα ποιότητα στην ε, απασχόληση, συνθήκες εργασίας, περιφερειακές διαφορές, ε, θα ενώσουν τις προσπάθειές τους οι μη προνομιούχοι και για να μπορέσουμε τώρα να δούμε τι μορφές μπορεί να πάρει αυτό το αριθμιστικό πλαίσιο. Έχουμε διάφορα κριτήρια, κάναμε μια συγκριτική ανάλυση και προτείναμε τέσσερις διαφορετικές επιλογές πολιτικής. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφαλεία δικαίου, προσαρμογή, δυνατότητα προσαρμογή του δικαίου σε σχέση με την ε, αποτελεσματικότητα και την αποδοχή. Το βασικό σενάριο θεωρούμε ότι είναι ότι θα πρέπει να μείνει ως έχει το σημερινό δίκαιο, δεν χρειάζεται κάποιο είδους προσαρμογή. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Για... Ε, όμως δεν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν δεν θα υπάρξει πολύ ε, αποτελεσματικότητα, ούτε θα άρει την απουσία ασφαλείας δικαίου. Ναι, μπορεί να υπάρξει μια οδηγία για μια μίνιμουμ εναρμόνιση. Να δούμε ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει μια τέτοια επιχείρηση. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Ούτε αυτό μας φαίνεται τόσο αποτελεσματικό σενάριο, γιατί θα πρέπει όλα τα κρατημέλη στην εθνική τους νομοθεσία να ενσωματώσουν τουλάχιστον μια νομική μορφή για αυτές τις επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει να βελτιωθούν όμως τα του συντονισμού των κρατών μελών. Θα πρέπει βέβαια να αλλάξει κάθε νομή τάξη για το τι θα χρειάζεται από κάθε τέτοια επιχείρηση για να αναγνωριστεί. Πάντως, ένα γενικό πλαίσιο δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά κάθε μιας τέτοιας επιχείρησης. Δεν θα αποτελεί κίνητρο για να πιάσουν το μήνυμα οι καταναλωτές για όσα παράγουν αυτές τις επιχειρήσεις. Ούτε θα τις προβάλλει τρίτη επιλογή. Ένα νέο σύστημα τικετοθεσίας και πιστοποίησης φαίνεται ότι είναι η πιο εξισορροπημένη λύση μεταξύ ασφαλείας δικαίου και ευελιξίας. Θα υπάρχει η maximum ευελιξία για τους επιχειρηματίες. Θα μπορούν να επιλέξουν ποια νομική μορφή ταιριάζει στα όσα χρειάζονται. Τα υπάρχοντα νομικά πρόσωπα θα συνήθως λειτουργούν και δεν θα χάσουν οι υπάρχουσες, μάλλον θα μπορούν να αλλάξουν νομική μορφή υπάρχουσες επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται η διάλυσή τους. Έτσι επίσης θα έχουμε κάποια εξοικονόμηση εξόδων. Δεν θα χρειάζεται να καταχωρηθούν σε κάθε κράτος μέλος για να αναγνωριστούν. θα είναι διακριτή η θέση του σε σχέση με άλλε εταιρείε, θα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προ επενδυτέ και καταναλωτέ. Με την ετικετοθεσία και την πιστοποίηση θα είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και θα υπάρξει και περισσότερη εμπιστοσύνη. Τέλος. Η προσθήκη κάποιας νομικής μορφής υπερεθνικής δεν θα δώσει πολύ ευελιξία στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για έναν τομέα καινοτόμο που τώρα αναπτύσσεται. Επίσης, από πολιτικής πλευράς δεν θα είναι τόσο αποδεκτό ένα τέτοιο μοντέλο. Εν κατακλείδη. Πολλές φορές η νομοθεσία έχει περιορισμένα αποτελέσματα χωρίς να υπάρχουν συνοδευτικές πολιτικές. Μπορεί να υπάρχει αναγνώριση αυτών των εταιριών από ένα ενωσιακό πλαίσιο, αλλά χρειάζεται επίσης μία σειρά δράσεων και σε εθνικό επίπεδο και σε κοινοτικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Προτείνω τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή το επόμενο σημείο αφορά το ίδιο θέμα. Είναι η εξέταση ενός σχεδίου έκθεσης ε, για, τις, ε, για το καταστατικό ε, των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Να συνενώσουμε τα δύο σημεία, να δώσουμε τώρα το λόγο στον εισηγητή και να κάνουμε μία συζήτηση και για τα δύο σημεία. Ο κύριος Μαστάλκα, λοιπόν, εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισχύτρια για την παρουσίαση. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για όλους μας. Υπογράμμισε τα σημαντικότερα προβλήματα και ζητήματα που, μας, που αποτελούν τροχοπέδι στη χρήση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων περισσότερο. Στη συνέχεια θα ήθελα να εστιαστώ στα τελευταία δύο ζητήματα που ανέφερε η προλαλή Η πρόταση για μια υπερεθνική νομική μορφή, όπως υπόθηκε, μου φαίνεται μη αποδεκτή από πολιτική άποψη αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να υπάρξει πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ε, θα μπορούσε να έχει άμεση εφαρμογή θα ήταν ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης, ε, κάτι που θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις ε, να αλλάξουν μορφή καταστατικού. Και έχετε δίκιο, ναι, πρέπει να εντείνουμε την ευαισθητοποίηση στο θέμα των επιχειρήσεων αυτών. Διότι τι άλλο στην Τσεχική Δημοκρατία, που είναι και η χώρα που γνωρίζω καλύτερα, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για την ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων. Ε, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το βελτιώσουμε. Έχω μία ερώτηση προς την ε, εισηγήτρια. Ε, ποιες χώρες δεν έχουν νομική μορφή για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ενδεχομένω μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό αργότερα, αφού κάνω εγώ την παρουσίαση του δικού μου εγγράφου. Κυρίε και κύριοι, Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το δικό μου σχέδιο έκθεσης ε, για τις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και το σχετικό καταστατικό. Ε, η έκθεσή μου εγώ ήθελα να ε, διακρίνεται από αισιοδοξία, από τα θετικά χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να τύχει ευρείας υποστηρίξης. Εδώ μιλάμε για πάνω από 40 εκατομμύρια απασχολούμενους, ε, τεράστιο ποσοστό ε, των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση έδειξε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα ε, το επέστησαν οι άνθρωποι από μειονεκτούσε κατηγορίε χαμηλών προσόντων, με αναπηρίε κτλ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ε, περιβάλλον ε, ευνοϊκό για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Γιατί, διότι δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ε, για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική καινοτομία. Ως εισηγητής της Επιτροπής Γιούρη, εγώ κλήθηκα να παρουσιάσω μια λύση ή λύσεις για το καταστατικό κοινωνικών και αλληλεγγύων επιχειρήσεων. Είχαμε μια δημόσια ακρόαση, εντατικές συζητήσεις με πολλούς ειδικού. και όλα αυτά με βοήθησαν να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι προς το παρόν είναι αδύνατο να, να απαιτήσουμε ομοιόμορφη νομική μορφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τέτοιες εταιρείες. Το λέω αυτό βάσει της δικής μου εμπειρίας με τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που έτυχε απόρριψης. Επίσης υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ε, στον τρόπο που ρυθμίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Τεράστια ποικιλομορφία οργανωτικών μορφών. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες νομικές απαιτήσει ε, κοινέ για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις όπως και αν αυτές ε, έχουν ε, συσταθεί και καταχωρηθεί. Ε, γι' αυτό τον λόγο προτείνω να εισάγουμε την επισήμανση, μια ευρωπαϊκή κοινωνική επισήμανση, η οποία θα είναι προαιρετική. Δηλαδή θα μπορεί να τοποθετηθεί εφόσον το ζητήσουν οι κοινωνικέ επιχειρήσεις. οποίο όμως χρησιμοποιεί αυτή την επισήμανση θα απολάβει τον ωφελόν του σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα μπορεί δηλαδή να μεταφερθεί ε, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Θα μπορεί να διευκολύνει τη χρηματοδότηση, ε, την διεξαγωγή διαγωνισμών, διότι θα είναι ευκολότερος ε, ο εντοπισμός ε, αυτών των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα εντό εισαγωγικών θα πρέπει να δίδεται σε επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό αναφερθήκε ήδη από την κυρία Τύριον. Θα αναφερόμαστε δηλαδή εδώ σε επιχειρήσεις που εργάζονται για το κοινό καλό. Επιχειρήσεις που λειτουργούν ε, δημοκρατικά. Εγώ σε αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, επισυνάπτω και ένα παράρτημα όπου μπορείτε να βρείτε και άλλες συστάσεις. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πετύχω είναι το εξής Θέλω οι κοινωνικές ε, ε, επιχειρήσεις να είναι προστατευμένες από την απάτη. Θέλω να καταλήξουμε σε μια κατάσταση την οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν όλες οι ομάδες. Οι προθεσμοί για τις τροπολογίες είναι 12 Ιανουαρίου του 2018. Κάποιοι συναδέλφοι από άλλες επιτροπές ε, ωστόσο μπορεί μπορεί να ψηφίσουν το Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα σημειωθεί καθυστέρηση και στη δική μας Επιτροπή. Αναμένουμε ψηφοφορία στη δική μας Επιτροπή το Μάιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Ρέγνερ. Ε, thank Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εκπροσωπώ τη Βυρζινή Ροζιέρ που δεν μπόρεσε να έρθει. Ομιλώ λοιπόν εκ μέρους της. Η Βυρζινή θα ήθελε να ευχαριστήσω τον κύριο Μαστάλικα για την πολύ καλή δουλειά του μέχρι τώρα. Σημερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειές του. Υπάρχει απουσία συνειδητοποίηση ως προς το ρόλο και τα αποτελέσματα της ε, κοινωνικής οικονομίας στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη ε, ποικιλία νομικών μορφών και ως εκ τούτου αυτό που βλέπουμε, αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει ο, ένας κοινό ορισμός και αντίληψη τι είναι η κοινωνική επιχείρηση, η επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας όπως άλλωστε προσπαθεί να εξηγήσει με την ερευνητική αυτή δουλειά ο κύριος Μασταλκαγή. Η κυρία Ρόζιερ πιστεύει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προαχθεί αυτό το τμήμα της οικονομίας, 25.000 οι επιχειρήσεις, 45 εκατομμύρια οι εργαζόμενοι. Επομένως πρόκειται για έναν τομέα που πραγματικά αξίζει να διερευνήσουμε περαιτέρω και να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό επίσης είναι να, να υιοθετηθεί ένας κοινό ε, ε, ορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια στην εσωτερική αγορά να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ή να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες της κοινή αγοράς της βασικής κοινωνικής επιχείρησης κατά τρόπον ώστε να έχουν νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πρόταση ε, είναι ρεαλιστική η κυρία Ροζιέ θεωρεί ως εκ τούτου ότι αυτή η ιδέα μιας σήμανσης που θα μπορούσε να στηρίζεται στο αντικείμενο και όχι τόσο στη νομική μορφή στον τύπο δηλαδή της επιχείρησης έχει πολύ μεγάλη σημασία δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο κάνει σαφή διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών φορέων ε, που δεν έχουν όμως σημασία για την κοινωνική οικονομία. Η κυρία Ρόζιερ πιστεύει ότι πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες να ξεπεράσουμε αυτή την βασική δυσκολία με την εισαγωγή ενδεχομένως μιας τρίτης κατηγορίας που έχει να κάνει με την χαμηλή κερδοφορία ε, επίσης η Βυρσινή πιστεύει ότι θα πρέπει να καταγραφούν οι εξελίξεις, ε, οι εξελίξεις της συνεργατικής λεγόμενης οικονομίας καθώς ε, σε μεγάλο βαθμό διεκδικεί θέση στην κοινωνική οικονομία και ενώ υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες που ανοίγουν με το ψηφιακό περιβάλλον και τη συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων που μπορούν να έχουν σαφή ε, ωφέλη για την κοινωνία. Πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όμως και να μην περιλάβουμε όλες τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας μόνο και μόνο επειδή ε, το δηλώνουν. Ε, αυτές είναι οι ιδέες της και παρακαλώ να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ Ράγεφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μαστάλκα. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί, να επιτύχει τους στόχους της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις αρχές βέβαια της αναλογικότητας και της υποκουρικότητα, χωρίς να απαιτείται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Πάντως, έχω κάποιες ερωτήσεις και συγκεκριμένα νομική βάση. Ποια είναι η νομική βάση, παρακαλώ. Η δική σας επιλογή είναι αυτή του άρθρου 50, που επιτρέπει την εγκαθίδρυση μιας νέας ε, νομικής μορφής. Αλλά δεν είναι αυτό ο στόχος μας, έτσι δεν είναι. Δεύτερον, με βάση τις εκθέσεις που πρέπει να δημοσιεύουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Αναφέρετε εσείς διάφορες παραμέτρους, μέσα στις οποίες καταλέγονται και οι μισθοί. Ναι, έστω να υπάρξει διαφάνεια αλλά δεν νομίζετε ότι ε, η δημοσίευση των αμοιβών, εάν βέβαια υπάρχουν και προβλέπονται αμοιβέ, θα δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ε, ανώνυμες εταιρείες, καταμετοχές ούτε με εκθέσεις ανακράτος. Επίσης για το παράρτημα αναφέρεται έναν ε, κατάλογο που θα μπορούσε να καταρτιστεί. Κατάλογο των διαφόρων νομικών ε, μορφών που θα μπορούσαν να ε, λάβουν κοινωνικό σήμα. Μα αυτές είναι επιχειρήσεις είτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε περιορισμένης κερδοφορίας. Τι μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος κατάλογος ή μη μόνον πρόσθετο ε, γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις απαντήσεις βέβαια και προσβλέπω στη συνεργασία. Παρακαλώ. Ε, ναι, πιστεύω ότι η βασική ιδέα του συναδέλφου Μαστάλκα, η κυρία Χάουτα, αλλά στην εξασφάλιση μιας ε, ε, σήμανσης των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι μια πολύ καλή ιδέα δεδομένη της απουσίας ομοιομορφίας ε, ως προς τις ε, νομικές μορφές των 28 κρατών μελών είναι καλή η προσέγγιση, μια προσέγγιση εναρμόνισης. Άλλωστε η κυρία Ρέγνερ εκ μέρου και της κυρίας Ροζιέ ανέφερε ότι χρειάζεται ένας κοινό ορισμός, ένας ορισμός ο οποίος θα καθοδηγεί και τα κριτήρια. Και αυτή η κατηγορία, η τρίτη κατηγορία που προτείνεται ε, για χώρες χαμηλής κερδοφορίας δεν είναι κακή Ίσως θα είναι καλό να την ε, εξετάσουμε. Μπορούμε να δούμε και την ε, απόδοση της επένδυσης ή ε, τον αντίκτυπο επενδύσεων ως όρο γιατί φερειπίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες ή σε, μεγάλο, σε βαθμό μεγάλης μεταποίησης, ψηλής μεταποίησης μπορούμε να δούμε τον παράγοντα της, του αντικτύπου της επένδυσης για τις ε, επιχειρήσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη βεβαίως ε, είναι προσιλωμένα στην υλοποίηση του θεματολογίου 2020 με τους στόχους της ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό να το αγνοήσουμε και ένας τρόπος να το πράξουμε είναι βεβαίως να ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι επιχειρήσεις της ε, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Γαλλία αλλά και γενικότερα την Ευρώπη διαδραματίζουν ε, ε, ρόλο σημαντικό και πάνω απ' όλα μας επιτρέπουν αν όχι να συγκρατήσουμε τον καπιταλισμό, πάντως να περιορίσουμε την σκληρότητα του. Ε, βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων στην Ευρώπη, κάθε χώρα έχει την ιδιωτερότητά της. Ίσως θα ήταν καλό να κοιτάξουμε πέραν ε, των ε, πλεονεκτημάτων που είναι, ε, μας βρίσκουν όλους σύμφωνους, να κοιτάξουμε να μην πιέσουμε προς ε, συγκεκριμένες λύσεις, να μην επιβάλλουμε συγκεκριμένες λύσεις. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση θα πρέπει να βρούμε τα κοινά χαρακτηριστικά των αλληλέγγυων και κοινωνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο η πρώτη διαπίστωση του συναδέλφου μας στα ΑΛΚΑ ε, είναι ακριβώς ότι τα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ αβέβαια και ασαφή και άρα χρειάζεται πολλή δουλειά για τον προσδιορισμό του. Χαρακτηριστικό υπαριθμών 3 παραδείγματι που αναφέρει επιχειρήσεις οι οποίες ε, για τον χρήστη και το προσωπικό ε, εξυπηρετούν σκοπούς ε, γενικού συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος. Επίσης χαρακτηριστικά αυτόνομα, τον, αυτόνομη δράση σε σχέση με τις κρατικές Αρχέ, Αυτονομία όμως και ανεξαρτησία που αναφέρεται στο κείμενο δεν εξυπηρετεί του ίδιου, δεν εκφράζει τις ίδιες έννοιε και γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατό να βάλουμε αυτήν την ευρωπαϊκή σήμανση που μπορεί να φαίνεται ανώδυνη, αλλά μιλήσουμε ότι θα συνοδεύεται και από έναν μηχανισμό ε, εποπτείας ευρωπαϊκό, δηλαδή νέα ανάμειξη της γραφειοκρατίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους εγώ προτείνω να αφήσετε ήσυχε τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Θα πάνε όλα πολύ καλύτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Αν θέλει η κυρία από το ΙΠΕΡΕΣ μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του εισηγητού. Ναι, ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ρωτήθηκε ποια κρατημέλη δεν έχουν νομοθετική πρόβλεψη. Δεν προβλέπουν κάποια νομική μορφή, δεν προβλέπουν κάποιο νομικό καθεστώς για αυτές τις εταιρείες Καμιά φορά υπάρχουν κάποιε συνδευτικέ πολιτικέ, αλλά είναι η Αυστρία, η Κύπρο, η Εστονία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Λετωνία. Κάτω χώρες, αλλά και η Σουηδία. Thank you very much. So... Ευχαριστούμε, λοιπόν Πρόεδρος. Σας επαναλαμβάνω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 12η Ιανουαρίου. Την μεσημβρία. Κύριε Μαστάλκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την αδειά σα. Να μην σχολιάσω σε όλα αυτά τα τόσο εμπνευσμένα που ακούσαμε. Απλώς χαίρομαι που θετικά βλέπουν το κείμενό μου οι συνάδελφοι. Και ένα από τα πιο σημαντικά που ακούστηκαν ήταν το τι νομική μορφή προτείνω εγώ να προτιμηθεί. Και ποια νομική βάση το 50 λέω εγώ, το άρθρο 50 που καλύπτει και τις εταιρείες με κερδοσκοπικό σκοπό και τις λοιπές. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη νομική βάση. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσίευση, νομίζω ότι αυτό μπορεί να ρυθμιστεί στην αιτιολογική έκθεση. Και επίσης συμφωνώ με όσο είπε η κυρία Χάουταλα. Δηλαδή, να προσέξουμε περισσότερο τις ε, εταιρείε που έχουν περιορισμένα κέρδη. Έχουν αυτές μεγάλες δυνατότητες. Περιμένω την σχετική τροπολογία σας κύριε Χάουταλα, θα βοηθούσε πολύ. Τώρα για τον κύριο Λεμπρετό. Ίσως είναι όλα τέλεια στη χώρα σας, γιατί έτσι μας τα περιγράψατε πάντως. Εγώ έχω να σας πω ότι οι εταιρείε που θέλουν να πετύχουν περισσότερα σε αυτό τον τομέα θέλουν να μπορούν να λειτουργήσουν διασυνοριακά. Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα και η φραγμή. Άρα μπορεί να βοηθήσει και η Επιτροπή και το Κοινοβουλίο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω γραφειοκρατία. Είναι φιλόδοξες αυτέ οι εταιρείε. Θέλουν να φτάσουν ψηλά. Χρειάζονται την διασυνορική συνεργασία. Θέλουν να γίνουν πιο γνωστές. Θέλουν περισσότερη ομοιογένεια στην ε, νομική ρύθμιση, στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που μα είπε η κυρία Ρέγνερ και νομίζω ότι θα βοηθηθεί και η υπόθεση. Ε, thank you Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο. Επομένως μπορούμε να ολοκληρώσουμε με αυτά τα δύο σημεία τη μέσα διάταξη και πάμε στο σημείο υπερθυμών 7. Έχουμε τώρα τη συζήτηση των ε, τροπολογιών για την προληπτική αναδιάρθρωση, δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για αύξηση αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάρθρωση άφερη και απαλλαγής. Τον ρόλο έχει η κυρία Αγγελικά Νίμπλερ που είναι η συγγήτριά μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ε, προτείνω μια επισκόπηση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιό μου, ευχαριστώντας βεβαίως πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους. 300 περίπου είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και έτσι αποδεικνύεται και το ενδιαφέρον στο θέμα της αναδιάρθρωσης και βέβαια των μέτρων της ε, πτώχευσης και της κάλυψης των ε, πιστωτών. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως να καταθέσουμε και τις συμβαστικές τροπολογίες συν ε, το χρόνο. Ξεκινώ με τις πολυάριθμες τροπολογίες που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις και συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ιδιαίτερη θέση τους. Πολύ σωστό αυτό, στην πρώτη ακρόαση άλλωστε για το θέμα αυτό και εξ αρχής υπογραμμίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως μάλιστα να είναι απαραίτητο να ε, θεσπιστούν ειδικοί κανόνες, ε, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να, προ, να προβλέπει ιδιαιτέρως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια οδηγία. Ε, όλα αυτά που βεβαίως περιμένω και από την ε, παρούσα εδώ σήμερα Επιτροπή να μας δώσει κάποιες ιδέες ώστε να έχουμε, γιατί βλέπω ότι είναι σαφέστατη η συμφωνία για μια ιδιαίτερη υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης βλέπω από τις ε, τροπολογίες που έχουν κατεθεί ε, πως φαίνεται πολλοί συνάδελφοι να θεωρούν ότι η διαδικασία της αναδιάρθρωσης χρειάζεται καθαριστή. Τι ρόλο πρέπει να έχει αυτός, από ποιο σημείο πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία, με ποιο τρόπο. Αυτά είναι λεπτομέρειε που μπορούν να διευκρινιστούν, αλλά πάντω βλέπω ότι γενικά την χάνει υποστήριξη σε αυτή η πρόταση. Επίσης, ε, στην διαδικασία της αναδιάρθρωσης ή ε, τα μέτρα αναβολής μεταξύ 70 ημερών και 6 μηνών με μέγιστο τους, τις 100 ημέρες τους 18 μήνες είναι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί μέσα των τροπολογιών. Κάπου θα τις συζητήσουμε τους ή άλλως, κάπου στα μισά θα βρούμε μια καλή λύση με βέβαιη. Τροπολογίες επίσης προτείνουν μια διαδικασία ε, που θα καλύπτει και φυσικά πρόσωπα εγώ πιστεύω ότι αυτό, και θα μα πει και η Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να επαφεθεί στα ίδια τα κράτη-μέλη αυτή η επιλογή. Αλλά κάποιοι συνάδελφοι με τις τροπολογίες προτείνουν ε, δεσμευτική την κάλυψη και των φυσικών προσώπων. δεσμευτική για τα κράτη-μέλη δηλαδή τη συμπερίληψη των φυσικών προσώπων. Θα το δούμε όμω, θα βρούμε μία λύση. Η 178 τροπολογία επίση αναφέρεται σε πολύ μικρέ επιχειρήσει και επιχειρηματίε οι οποίοι αναλαμβάνουν ευθύνη με την προσωπική τους ε, περιουσία. Πολύ σημαντικό το θέμα, ένα από τα κεντρικά ζητήματα που δεν ξέρω πώς θα λύσουμε, αλλά οπωσδήποτε θα μας απασχολεί στις περαιτέρω συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή και βέβαια και τις συνομιλίες ε, με τους σκιώδεις εισηγητές. Και υπάρχει και το θέμα βεβαίως που πρέπει επίσης να συζητήσουμε με τους και του ηγητές των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έχουν κατευθεί πολλέ τροπολογίε. Οι προληπτικές διαδικασίες ε, εκαθάριση αναδιάρθρωσης πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή και διαφύλαξη των εργαζομένων, ε, συμμετοχή των εργαζομένων και διαφύλαξη των δικαιωμάτων του τα δικαιώματα των εργαζομένων παραμένουν, δεν φύγονται με βάση την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν δημιουργούνται και νέα δικαιώματα εργαζομένων με βάση την υφιστάμενη ε, διαδικασία. Σημαντικό πάντω είναι να μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στι διαδικασίε αυτέ τη αναδιάρθρωση. Πολλέ είναι που έχουν κατευθεί και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο ώστε με ηρεμία να μελετήσουμε τι έχει νόημα να συμπεριλάβουμε και να προβλέψουμε για αυτέ ε, τι δυνατότητε συμμετοχή των εργαζομένων, έτσι ώστε και η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά και να μην αποκλείονται οι εργαζόμενοι, γιατί χωρί εργαζομένου δεν μπορεί να υπάρχει η λειτουργία τη επιχείρηση. στην αναδιάρθρωση για λόγου οικονομικού είναι μια άλλη διαφορετική υπόθεση, δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε με ε, ανα αναδιάρθρωση χρεών κτλ. Και, και όταν πρέπει κανεί να στραφεί στι αγορέ για να βρει λύσει για χρηματοδότηση επιχείρησή του υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, προσεγγίσει οπωσδήποτε. Εγώ θα υποστηρίξω λύσεις λογικές για τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Και τελευταία παρατήρηση. Ε, για τις ε, τροπολογίες που έχουν κατεθεί από πότε και ποιο χρονικό σημείο έχουμε να κάνουμε με την οριστική πλέον πτώχευση, ε, οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους έχουν μιλήσει για μια προθεσμία η οποία θα ανέρχεται από το πολύ, από το ελάχιστο 3 μέχρι μέγιστο 5 έτη. Το θέμα δεν νομίζω ότι θα κρυθεί βέβαια στην ε, προθεσμία και την διάρκεια της διαδικασίας της πτώχευσης. Οπωσδήποτε θα βρούμε κάποια λογική λύση. Ε, για μένα καθοριστικό είναι να έχουμε μια συνολική λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική. Ε, σε μια πρώτη ανάλυση αγαπητοί συνάδελφοι αυτό έχω να πω ε, περιγράφοντας μόνο τα θέματα που μας απασχόλησαν ε, σε σχέση με το ζήτημα και προσκαλώ εννοείται τους συναδέλφους σε μια, σύνοδο, σε μια διάσκεψη με τους σκιώδεις ώστε να συζητήσουμε, να ομαδοποιήσουμε τις ε, προτάσεις ή θεματολογικά τουλάχιστον τα σημεία που έχουν ε, αναφερθεί και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέγνερ. Πάλι σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να σας μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Κοφεράτη που είναι ο σκιώδης Σύμφωνα με τις τροπολογίες του Πάντω τώρα θα σα πω τη δική του γνώμη με την οποία συμφωνώ απολύτω. Είναι 100% απαραίτητο να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα αναγκαία μέσα τόσο να έχουμε αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων πριν αρχίσει η κανονική διαδικασία ε, της Οπότε θα πρέπει να σωθούν οι ε, αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην οικονομία στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποια ευαισθησία, να προσέξουμε πώς ρυθμίζουμε αυτά τα θέματα. Οπότε και εμείς συμφωνούμε 100% με τα προτείνει η Αγγέλικα Νίμπλερ. Τώρα, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλο των εργαζομένων για αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία τη αναδιάρθρωση και ιδιαίτερω όσον αφορά την ενημέρωση και την έγκαιρη εμπλοκή του. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και αφορά το τι θα γίνει με την μέλουσα πιθανή αφαιρεγγιότητα. Και εδώ συμφωνώ με την Επίση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξουν αποφάσει που να οδηγήσουν σε ουσιώδει μεταβολέ όσον αφορά την οργάνωση τη ε, δουλειά ή τη σχέση εταιρεία. Γιατί κάποιοι οποίοι θίγονται από αυτή την αναδιάρθρωση θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για αυτέ τι αποφάσει και να, έτσι να, να, να ανακλείσει το deal, το, το, το πλάνο τέλο πάντων Οπότε εμεί αυτό το οποίο θέλουμε να ισχύσει το ότι δεν όλοι οι πιστωτέ το ίδιο θα πρέπει να προστατευτούν περισσότερο οι πιο αδύναμοι από τους πιστωτέ. Κάτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν διαφορετικέ κατηγορίε πιστωτών και θα πρέπει οι αξιώσεις αντίστοιχα να έχουν κάποια κατάταξη. Οι πιο δυναμικοί από τους πιστωτέ βέβαια είναι οι εργαζόμενοι. Τα κρατημέλη θα πρέπει να νομοθετήσουν ακριβώς τον διαχωρισμό των εργαζομένων και θα πρέπει να είναι προνομιούχα η αξίωσή του. Ισχύει αυτό σε κάποια κράτη-μέλη. Ή είναι αυτό η συνήθις συνηθες ρυθμιση φυσιολογική επιλογή. Αλλά αυτό θα πρέπει να ισχύσει και πανευρωπαϊκά. Τώρα συμφωνούμε με αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα υπάρχει, να υπάρχει μια εύλογη περίοδο ε, μεταβατική, περίοδο παγώματο στην αναδιάρθρωση, αλλά θα πρέπει να αυτό να μην ε, έχει επιπτώσεις στην αμοιβή των εργαζομένων. Οπότε θα πρέπει εδώ να υπάρξει πιο στεγανή ρύθμιση εξασφάλισης. Τέλος ο ρόλος των προσώπων καθέκαστων και των οικογενειών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει φυσικά τις επιχειρήσεις. Ακόμα σε νομοθετικό επίπεδο προσπαθούμε να δούμε πώς θα απορροφηθούν οι συνέπειες από αυτή την κρίση. Και αυτό φορά και τις οικογένειες Άρα τι θα πρέπει να είναι η την που θα περάσουν οι ρυθμίσει τη Επιτροπή. Υπάρχουν βέβαια διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών στο νομοθετικό επίπεδο, οπότε δεν μπορούμε απλώς να κάνουμε μία αυτόματη μεταφορά για τα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο. Πάντως κάτι θα πρέπει να γίνει. Οπότε θα ήθελα αυτό να σας υπενθυμίσω εγώ και ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρίν Μαρίν Πίντου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ ε, την εισηγήτρια. Συμφωνώ με τις ανησυχίες και τους στόχους της. Καταφέραμε και εμείς να συμβάλλουμε με κάποιες τροπολογίες. Ήθελα να ειδοποιήσω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αντίφασης δυνητικός. Πρέπει να τον προλάβουμε. Εδώ μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, μπορεί να χρειαστεί να ε, εφαρμόσουν μια τέτοια διαδικασία δεύτερης ευκαιρίας ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν, προσπαθούν να αποφύγουν ε, την αφαιρεγκαιότητα ε, επιχειρήσεων οι οποίες θα ήταν βιώσιμες ε, αν είχα μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό συμβαίνει ή απλά προσπαθούμε να παρατείνουμε τεχνητά τη ζωή μιας επιχείρησης που είναι επιβλαβής για την αγορά και που θα συνεχίσει να είναι επιβλαβής για την αγορά. Αυτού του ο μηχανισμός απαιτεί πολύ αυστηρή και λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης. Αυτό διότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να καταστραφεί μια επιχείρηση παρά να παρατείνει τεχνητά τη ζωή της ε, και να συνεχίσει να δημιουργεί ζημία στους πιστωτές της ε, λόγω μη πληρωμών κτλ. Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο και πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνουμε στους άνθρωπους μια δεύτερη ευκαιρία. Αφού όμω ε, πρώτα έχουμε ελέγξει κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί η κατάσταση. Συμφωνώ με τις απόψεις του κυρίου Κοφεράτη. Πρέπει να ακούσουμε και τις φωνές των εργαζομένων σε αυτές τις διαδικασίες, διότι είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ε, όσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις και την ε, συνέχιση της ζωής τους. Θα πρέπει λοιπόν να τους προφυλάσσουμε ακόμα και στην περίπτωση όπου η σωστή λύση για μια εταιρεία είναι να διαλυθεί. Ένα κομμάτι των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσης που αντιστοιχούν στα συνταξιδοτικά ταμεία θα πρέπει να διατηρηθεί. Να μην είναι κομμάτι της αφαιρεγγιότητας, διότι πρόκειται για ε, συνεισφορές ε, των εργαζομένων για τις συντάξεις τους. Αυτές θα πρέπει να χαιρούν πρόσθετης προστασίας και φυσικά θα πρέπει να ακούμε και τις φωνές των εργαζομένων, ειδικότερα των εκπροσώπων τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εμπειρία και την νομική κατάρτιση και ιδιότητα τέτοια ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο την κυρία Νίμπλερ για αυτό το σχέδιο, οδηγίας, ε, για το σχέδιο για την οδηγία η οποία προβλέπει ε, την προαιρετική αίτηση ενός ε, οφειλέτη για αναστολή των διαδικασιών κατά το ατόμο του. Αυτό αφορά και τι διαπραγματεύσει για την αναδιάρθρωση. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα επιχειρηματία που ζητά να ξεκινήσει μια διαδικασία αναδιάρθρωση δεν μπορεί να είναι βέβαιο για την ανάκληση των ε, ατομικών διώξεων. Ε, ανάκληση που θα του έδινε λίγο χρόνο να αναπνεύσει, λίγο χρόνο να καταλήξει κάποια συμφωνία με τους ε, πιστωτές του αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόβλημα ε, και με τους πιστωτές διότι το κριτήριο της ανάκλησης μη ανάκλησης των ε, ατομικών διώξεων δεν είναι σαφές. Επίσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος. Αυτό θα δημιουργούσε και πρόβλημα στην επίτευξη της επιθυμητής εναρμόνισης. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προβλέψουμε ότι η δικαστική απόφαση ανάκλησης της ε, ε, ε, δικαστική απόφαση αναδιάρθρωσης θα οδηγεί σε ανάκληση των ατομικών διώξεων και στην εκκίνηση μιας διαδικασίας αφαιρεγγιότητας διότι Διαφορετικά μπορεί να είναι η όλη διαδικασία επιβλαβής για τις διαπραγματεύσεις αναδιάρθρωσης. Όσον αφορά τις προθεσμίες, ε, που χορηγούνται στον οφειλέτη σε περίπτωση αναστολής των διώξεων. Ε, η προθεσμία αυτή είναι δίμηνη. Σε περίπτωση που αποφασιστεί δικαστικά να παραταθεί αυτή η προθεσμία, παρατείνεται στου έξι μήνες. Ωστόσο, θεωρώ ότι η προθεσμία αυτή είναι πολύ μικρή. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιστεύω θα εμποδίσει την ε, αναδιάρθρωση. Θα ήθελα επίσης να προτείνω στα κράτη-μέλη να εισάγουν κανόνες ε, που θα αφορούν την αφαιρεγιότητα των πελατών ε, το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά την ανάκληση των διαόξεων κατά του οφηλέτη, όταν ε, έχει ξεκινήσει από μια δικαστική αρχή η διαδικασία αναδιάρθρωσης, θεωρώ ότι σκόπιμο θα ήταν να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα για τον πιστωτή να ζητήσει ακύρωση αυτής της ανάκλησης. Ελπίζω να υποστηρίξετε αγαπητοί συνάδελφοι τις τροπολογίες που υποβάλλω προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον κύριο Στάιν από την Γενική Διεύθυνση Τζάστα. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, πολύ σωστά. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτές τις έντονες συζητήσεις και τις πολυάριθμες τροπολογίες. Ενημερωτικά και θα το γνωρίζετε ήδη θα εξεταστεί αυτό το θέμα ε, στην συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνη ε, αύριο και τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η απέτηση βιωσιμότητας για την πρόσβαση στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ο μηχανισμός ε, αντίστροφου υπολογισμού και η απαλλαγή. Πολλά σημαντικά ζητήματα λοιπόν θα συζητηθούν στο Συμβούλιο και τα βρίσκουμε και στις τροπολογίες. Ας δούμε αυτά τα ζητήματα λοιπόν, διότι προέκυψαν εδώ στη συζήτηση και μετά θα απαντήσω σε κάποια ε, σε από τις άλλες παρατηρήσεις που ακούσαμε. Η βιωσιμότητα. Πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί για την ειδική περίπτωση μιας επιχείρησης που απαιτεί ε, προσφυγή σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης και έχουμε προτάσεις ε, για την πιθανότητα της, ανα... της ε, του να σωθεί από αυτό, για τη βιωσιμότητα. Πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε το ίδιο πράγμα εδώ, αλλά είναι δύσκολο να το ορίσουμε. Όλοι συμφωνούμε ότι μια επιχείρηση πρέπει να ασθενεί για να έχει πρόσβαση σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Αν είναι υγιής δεν χρειάζεται, αλλά μπορεί να ασθενεί τόσο πολύ που να είναι η διαφερέγγια και θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική ε, θεραπείας από αυτή την ασθένεια. Αυτό που ανέφερε λοιπόν ο κ. Πίντο για το κίνδυνο τεχνητής παράτασης της ζωής μιας επιχείρησης ε, δεν είναι καθόλου σκοπός αυτής της οδηγίας αυτός. Θέλουμε να γίνεται μια σαφή διάκριση για τι περιπτώσει όπου δεν υπάρχει ελπίδα και που θα περνούν από απλέ διαδικασίε αφαιρεγγιότητας και μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν προβλήματα αλλά όπου υπάρχει ελπίδα. Το θέμα είναι πώ το αποτυπώνει αυτό κανεί σε ένα νομοθετικό κείμενο. Εγώ διακρίνω κάποιον κίνδυνο αν προσπαθήσουμε να είμαστε υπερβολικά ακριβεί. Κάποιοι από αυτού του ορισμού δεν είμαι βέβαιος ε, η προστιθέμενη αξία ε, εμπεριέχουν. Επίση, δεν θέλουμε να γίνει υπερβολικά επαχθή η διαδικασία, διότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίε, αν καταλήξουν σε μια νομική μάχη προσπάθειας ερμηνεία των ορισμών και εκεί θα περιπλέκει η κατάσταση. Ε, πιστεύω ότι θα βρούμε συμφωνία. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτή τη φάση ότι υπάρχει ένα σημαντικό παράγον που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το ρόλο των πιστωτών. Μια επιχείρηση, αν είτε είναι πολύ υγιή ή πολύ ασθενή, οι πιστωτέ τη δεν θα είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν στη διαδικασία. Αιτιολογείται δηλαδή το επιθετικό σενάριο ότι αν επαρκής αριθμός πιστωτών θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη ε, διαδικασία βρισκόμαστε στην κρίζα ζώνη όπου μια ε, επιχείρηση δεν είναι ακόμη αφαιρέγγια αλλά αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ε, και βρίσκεται υπό την απειλή αφαιρεγγιότητας οπότε θέλουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για να καταφέρουμε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πρόταση Το Clamp Clampdown ε, το συζητήσαμε πολύ ε, για την κατηγοριοποίηση ουσιαστικά των ε, πιστωτών. Θα πρέπει να δούμε τι κατηγορίες θα υπάρχουν. Καταλαβαίνουμε τη λογική και αν υπάρχουν πολλές κατηγορίες είναι σαφές γιατί θα χρειαστεί κάποια υποστήριξη για να οριστούν σωστά αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ήδη το κείμενο δίνει ε, ευελιξία. Υπάρχει μια κατηγορία ω αφετηρία και μετά τα κράτη-μέλη επ' αυτού μπορούν να ρυθμίσουν και να κάνουν τι απαραίτητε τροποποίησει. Επίση πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το μόνο που προβλέπει η οδική ελάχιστη εναρμόνιση ε, είναι δύο κατηγορίε, ασφαλή και μη ασφαλή. Ε, και σε πολλά κράτη-μέλη ούτω ή δεν θα χρειαστεί να υπάρχουν περισσότερε από δύο κατηγορίε και αυτό καθιστά προβληματική την έννοια της ε, πλειοψηφίας των ε, ε, κατηγοριών, διότι η πλειοψηφία των δύο είναι δύο. Οπότε εκεί υπονομεύουμε ολόκληρη την έννοια της εξισορρόψης μεταξύ των κατηγοριών. Οπότε πρέπει να δούμε τι καταστάσεις θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πόσο διαφορετικές είναι αυτές και ποια θα είναι μια λογική λύση. Τώρα, για τις περιόδους απαλλαγής που αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια και από κάποιους άλλους συναδέλφους, όπως όλες οι προθεσμίες και αυτή υπόκειται σε συζήτηση. Απαιτείται συζήτηση για να βρούμε κάποια πολιτικά ορθή ισορροπία. Πρέπει να πω ότι ήδη η περίοδος απαλλαγής ε, που είχε συμφωθεί στο Συμβούλιο αρχικά ήταν τριετής. Ε, πριν από μερικά χρόνια είχε ληφθεί αυτή η απόφαση. Θα ξανακάνουμε τις συζητήσεις, αλλά το μόνο που έχω να πω στην παρούσα φάση είναι ότι θεωρούμε πως δεν έχει νόημα να υπάρχει ελάχιστη περίοδος. Αυτή είναι μια από τις προτάσεις μας, να έχουμε τουλάχιστον τρει διότι θέλουμε να πετυχαίνει η δεύτερη ε, ευκαιρία. Όταν λέμε ότι ο χρόνος απαλλαγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3, ενώ ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, 12. Ε, Οπότε έτσι να μην ε, συντελείται ποτέ πραγματική απαλλαγή. Θέλουμε να υπάρχει μια μέγιστη περίοδος λοιπόν και είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει σωστή ισορροπία με τα τρία έτη. Τώρα κάποιες άλλες παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα. Ε, διάρκεια παραμονής ε, αποτελεί χαρακτηριστικό κλειδί. Έχει δώσει μια επισκόπηση η συγγήτρια για το ευρύ φάσμα που βλέπουμε στις διάφορες τροπολογίες. Όταν κοιτάει κανείς όλες αυτές τις τροπολογίες αποκτά την αίσθηση ότι τελικά να μην έχουμε κάνει απόλυτο λάθος στην πρότασή μας ε, σε αυτή που υποβάλαμε αρχικά αλλά όπως είπα, όπως και για τα υπόλοιπα ζητήματα, είμαστε διατεθειμένοι να σας παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη. Τώρα, για κάποια από τα άλλα ζητήματα που αναφέρθηκαν στη συζήτηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ναι, αποτελούν προτεραιότητα για την Κομισιόν ε, και στην πρότασή της. Ε, γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες ε, διατάξεις ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, ε, το σχέδιο ε, αναδιάρθρωσης αναενότητες που μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κάνουμε συζητήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε όλο αυτό. Απλά θέλω να τονίσω εδώ, να το συνδέσω αυτό με κάποια άλλα ζητήματα που συζητάμε. Όταν λέμε για υποχρεωτική αφαιρεγγιότητα ε, ή το τεστ βιωσιμότητας. Όσο πιο απαιτητικοί γινόμαστε σε σχέση με αυτές τις απαιτήσει, τόσο ανεβαίνει το κόστος και η δυσκολία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν και το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα ε, της πρότασης. Τέλος, άλλες δύο παρατηρήσεις ή μία η οποία προκύπτει και σε κάποιες ε, τροπολογίες είναι πώς προστατεύουμε τα συμφέροντα των πιστωτών ε, και ειδικότερα των πιστωτών με ασφάλεια. Σε αυτούς ε, προσπαθούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο ή κάποια συγκεκριμένα προνόμια διασφαλίζοντάς τους, προστατεύοντάς τους από την όλη διαδικασία διότι επειδή έχουν αυτές τις ασφάλειες, πρέπει, τις εγγύησεις πρέπει να ε, τους αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί οι security creditors, ε, οι εγγυημένοι ε, πιστωτές, πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία, διότι είναι αδύνατο να γίνει σωστή αναδιάρθρωση χωρίς τη συμμετοχή τους. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν, θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και τις συνέπειες, διότι οι μη προστατευόμενοι πιστωτές και αυτοί πρέπει να έχουν ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια δίκαιη λύση για όλους να συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές για την αναδιάρθρωση. Τέλος, δύο λόγια για το ρόλο των εργαζομένων. Εμείς κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να πούμε ότι αυτό δεν θα προσβάλλει κανένα δικαίωμα εγγυημένο για τους εργαζομένους υπό εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι μόνες συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια πρόταση για τους εργαζομένους είναι ότι μπορεί να αποκτήσουν επιπλέον δικαίωματα, επιπλέον των όσων έχουν ήδη. Αν μια αναδιάρθρωση σημαίνει αλλαγή σε μια επιχειρία η οποία δυνάμει του διεθνούς δικαίωμα οδηγεί σε κάποια δικαιώματα απόφαση απόφασης, όλα αυτά φυσικά παραμένουν. Επιπροσθέτως όμως οι εργαζόμενοι ως ξεχωριστή κατηγορία αποκτούν και δικαιώματα ψήφου εφόσον το σχέδιο τους επηρεάζει. Εμείς πιστεύουμε ότι πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ουσιαστικά αποτελούν διευκρινήσεις ε, των δικαιωμάτων των οποίων θα απολαύουν ήδη οι εργαζόμενοι δυνάμει της απόφασης αυτής όπως το κατανοούμε εμείς. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι για περαιτέρω συζητήσεις ε, για να το διευκρινίσουμε καλύτερα στο κείμενο. Αλλά και εδώ θα ήθελα να ε, προειδοποιήσω ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τα όρια αυτής της πρότασης και αυτής της οδηγίας όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους δώσουμε μια προνομιούχο θέση ως πιστο, όπως τους πιστωτές γιατί εκεί παρεμβαίνουμε στα ε, προνόμια δυνάμει της νομοθεσίας περί αφαιρεγκαιριότητας. Ε, κάποιοι το κάνουν αυτό εργοδότες, παρέχουν τέτοια δικαιώματα στους εργαζομένους αλλά εμείς δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην ε, νομοθεσία περί αφαιρεγγιότητας γιατί εκεί μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση και περιπλέκεται ε, ε, κατά πολύ η κατάσταση και η συζήτηση. Δεν μπορούμε να παρεμβούμε στην ταξινόμηση των κατηγοριοποίηση ουσιαστικά των πιστωτών διότι αυτό είναι θέμα νομοθεσίες περί αφαιρεγγυρότητας. Οπότε πρέπει να έχουμε στο νου μας διαρκώς τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων εντός του πλαίσιου αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλει η κυρία Νίμπλερ να προσθέσει κάτι. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως τους συναδέλφους επί τη ευκαιρία για τις τοποθετήσεις και τα σχόλιά τους. Ε, είναι πολύ χρήσιμα. Και βεβαίως μπορούμε να συστήσουμε τα διάφορα θέματα που εθίγησαν και σήμερα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Στάινερ, ο εκπρόσωπος Επιτροπής, ε, σημειώνουμε και είναι σαφές σε όλους ότι δεν μιλούμε για τη διαδικασία της πτώχευσης. Μιλούμε για ένα μέρος, για ένα κομμάτι της διαδικασίας πριν από την πτώχευση, την προληπτική ε, αναδιάρθρωση, η οποία ακριβώς προσπαθεί να αποφεύγει και προσπαθούμε επίσης να μην αφήσουμε να ξεφύγει και να καλύψει και θέματα της πτώχευσης. Τα δικαιώματα των εργαζομένων καλύπτουν μεγάλο κομμάτι αυτής της έκθεσης. Εγώ προσωπικώς γνωρίζω αρκετά καλά το γερμανικό πτωχευτικό δίκαιο, αλλά δεν είμαι εξοικειωμένη με τα αντίστοιχα δίκαια των κρατών μελών. Γι' αυτό θέλω ε, να μου επισημάνετε αν υπάρχει κάτι το οποίο έχω παραβλέψει ε, και θα ήθελα με τον κατάλογο μου να μου επισημάνετε αν κάτι υπάρχει σχέση με τη διαδικασία πτώχευση στα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ή να προβλέψουμε. Κάτι που ενδεχομένω περιτεύει κιόλα. Θα ήταν σκόπιμο να μου δώσετε μια επισκόπηση και έτσι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η κάλυψη των θεμάτων. Προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συζητήσει. Ε, μαθαίνω ότι και η Βουλγαρική Προεδρία, αυτό προς τον συνάδελφο Ράτεφ, έχει δεσμευθεί να προωθήσει περαιτέρω το φάκελο αυτό. Και πιστεύω ότι ίσως καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 18 να κλείσουμε το θέμα τελείως, αλλά μια πρώτη ανάγνωση, εν πάση περιπτώσει κάποια βήματα πρόοδου θα ήταν καλό και για μας εδώ στην Επιτροπή νομικών υποθέσεων οπωσδήποτε ε, δεν θα επιβραδύνουμε εμείς τη διαδικασία ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στις καλύτερες δυνατές προθεσμίες ευχαριστώ πολύ σημείο 9 ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικτυακή και άλλες εξαποστάσεις πωλήσει προϊόντων με την κυρία Χάουταλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 31 Οκτωβρίου έδωσε την ε, τροποποιημένη της πρόταση για την νομοθετική αυτή πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όχι τόσο αναπάντεχο, μάλλον αναμενόμενο ήταν το ότι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής από τις διαγραμμικές και άλλες εξαποστάσεως αποστάσεως αγαθών ε, σε όλες τις πωλήσει. Πεδίο εφαρμογής λοιπόν και άρθρο 1 και άρα πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος. Δεν μιλούμε μόνο για ε, εξαποστάσεως αποστάσεως αλλά για κάθε τύπο πωλήσεων. Και ενδέχεται αυτό να οδηγήσει και σε απλοποίηση της υπόθεσης. Μπορούμε δηλαδή να δούμε εναρμονισμένους κανόνες μεταξύ διαγραμμικών και μη πωλήσεων, συμβάσεων πωλήσεων, πράγμα το οποίο έχει ε, τεράστια σημασία και βέβαια έχει και νόημα τόσο για τον ε, πολίτη όσο και για τον καταναλωτή. Αυτό που βλέπω πάντως εγώ με την... Ε, με συγχωρείτε αλλά το παρακάνατε με τη φασαρία πρόεδρε, μήπως μπορούν όσοι δεν ενδιαφέρονται... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, ό,τι θέματα έχετε να τα συζητείτε εκτός της αιθούσης. Ακόμα και οι κυρίες που βρίσκονται στην είσοδο παρακαλώ και που φαίνεται δεν με ακούνα γιατί φαίνεται ότι ακόμα μιλάνε. It's more quiet now, so I continue. So, um... Να σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ας συνεχίσω τώρα. Όταν λοιπόν κατέθεσε τον Ιούλιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της, δεν προξένησε πάρα πολύ συζήτηση ή σ' άλλο, πέραν του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που βέβαια είχαν τις αρμοδιότητες, αλλά έχει έρθει πια η στιγμή, πιστεύω, να ανοίξει το θέμα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και σε επίπεδο κρατών μελών και έχουμε να κάνουμε με μια ουσιαστική ανατροπή της νομοθεσίας ε, της σχετικής με την προστασία του καταναλώτη. Πρόκειται για ρηξικέλευτη κίνηση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα συμφέροντα που ενδεχομένως εδώ διακυβεύονται για να τα εξισορροπήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Το Συμβούλιο έχει αρχίσει επιτέλους να συζητεί την πρόταση με μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πριν από μια εβδομάδα αν δεν απατώμε. Προσεχής προβλέπεται μέσα στο μήνα και άρα και εμείς παρακολουθούμε κατά πόδα. Ε, η πρότασή μου συγκεκριμένα είναι η εξή. Μια και έχουμε δύο μια και έχουμε νέα τροποποιημένη πρόταση, θα ήταν καλό να ανοίξουμε τουλάχιστον ε, μια σύντομη προθεσμία για τροποποίηση ε, για νέες τροπολογίες συγκεκριμένα και αυτό γιατί, διότι έχουν αλλάξει και τα άρθρα αλλά και το προήμιο και έτσι μπορούμε να επιτρέψουμε περιορισμένης διάρκεια όπως είπα, παράταση της ε, προθεσμίας για τροπολογίες μέχρι τι 11 Δεκεμβρίου, γιατί βέβαια και αυτό το θέμα μας απασχολεί εδώ και καιρό. Θα αρκέσει λοιπόν η ε, προθεσμία στις 11 Δεκεμβρίου και επίσης ε, η γνωμοδότηση του άρθρου 54 προς την ΙΜΚΟ από τη δική μας την Επιτροπή δεν πρέπει να κατεθεί βεβαιασμένα τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν ένα περιθώριο για να εγείρουν παρατηρήσεις σχετικές με την επικουρικότητα έως τις 24 Δεκεμβρίου παραμονή Χριστουγέννων. Και άρα και εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό εξασφαλίζοντας, όπως είπα, μια σύντομη προθεσμία για περαιτέρω τροπολογίες για τα άρθρα του διατακτικού και του προημίου που έχουν ε, ε, αναδιατυπωθεί και συγκεκριμένα για να δώσω το πρόγραμμά μου προτείνεται στις ψηφοφορία στην Επιτροπή 25 Ιανουαρίου. Επομένως πριν από την προθεσμία των 8 εβδομάδων για τις ε, Παρατηρήσει επικουρικότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων και είναι δική μα αρμοδιότητα η επικουρικότητα όπω καταλαβαίνετε. Τέλο πάντων εμείς δεν θα έχουμε τελειώσει τη δουλειά μα μέχρι τότε. Ε, δεν θα με ξαφνιάσει να κατεθούν επιφυλάξει επικουρικότητα, διότι ουσιαστικά αυτό που ε, συζητούμε είναι το επίπεδο εναρμόνιση τη καταναλ... της ε, νομοθεσίας για τους καταναλωτές και βεβαίω υπάρχουν κράτη που έχουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας από ό,τι άλλα. και είναι πολλαπλές οι διαφορές και πολλά τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε σωστά και τη δική μας την ε, διαδικασία εδώ στο Κοινοβούλιο, ώστε στα τέλη Ιανουαρίου να ψηφιστεί και να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς που προγραμματίζει την ψηφοφορία της το Φεβρουάριο για να πάει στην Ολομέλεια το θέμα ε, την Άνοιξη αυτό και θα σας υπενθυμίσω πως πρόκειται για μια διαδικασία παράλληλη προς μια πιο ε, προχωρημένη ως προς την επεξεργασία της ε, οδηγία σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο. Σας είναι οικία φαντάζομαι. και εδώ έχουμε φτάσει σε επίπεδο διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αισθάνομαι πάντως μια κάποια ανακούφιση γιατί τη βαριά δουλειά σε σχέση με το ψηφιακό περιεχόμενο την έχουμε λίγο πολύ ολοκληρώσει και έτσι μπορούμε πια να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στα απτά προϊόντα. Θέλαμε, η αγαθά, θέλαμε βεβαίω να πάνε παράλληλα οι δύο οδηγίε, αλλά είναι καλό που έχει τελειώσει το μεγάλο κομμάτι του ψηφιακού περιεχομένου για να περάσουμε στι διαγραμμικέ και μη πωλήσει αγαθών, υλικών αγαθών. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Σκιώδης, ο Σκιώδης εκ μέρους του ΕΛΚΟ και ο Γκοργά μου ζήτησε να σας διαβάσω την παρέμβαση του για αυτή τη γνωμοδότηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Σκιώδης του ΕΛΚ για τη γνωμοδότηση αυτή που αφορά ορισμένες πτυχές ε, της ε, πώλησης ε, αγαθών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή μας. Είναι μια τεράστια πρόοδος για μια πιο ολοκληρωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω απόλυτα το κείμενο του αρθρού 21 που προσεγγίζει την οδηγία για κάποιες ε, πτυχές ε, πώλησης και εγγύησης ε, των καταναλωτών. Θα αποτελέσει πλήρη εναρμόνιση μεταξύ των πωλήσεων online και των πωλήσεων σε καταστήματα. Έτσι, έρουμε την, την, τα προβλήματα ασφάλειας δικαίου για τους εμπόρους και τους καταναλωτές και διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη μετάβαση στις διασυνοριακές πωλήσει οι εναρμονισμένοι κανόνες θα παρέχουν ίσους, ίσες συνθήκες για όλες τις επιχειρήσεις. Κάτι απαραίτητο για να παγιώσουμε μια λειτουργική εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους καταναλωτές η οδηγία αυτή όπως τροποποιείται θα διασφαλίσει ίσο επίπεδο προστασίας, νομικής προστασίας στις επιγραμμικές πωλήσει και τις πωλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, όσον αφορά τι επιγραμμικέ αγορέ. Θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά του τηρούνται εξίσου καλά. Αυτό θα έχει θετικά αποτελέσματα και για τι διασυνοριακέ πωλήσει. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει την προσθήκη των εμπορικών εγγύσεων ε, όσον αφορά τη διάρκεια ζωή, όπω προβλέπεται στο άρθρο 15. Σύμφωνα με μια μελέτη αντικτύπου, που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο ε, μια τέτοια εγγύηση θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως ε, για ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Αναμένω με ανυπομονησία την ε, συνεργασία με, τον με την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Αυτή τη φορά εκπροσωπώ την κυρία Γκέπχαρτ για το θέμα αυτό η ομάδα μας υποστηρίζει ανέκαθεν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής διαγραφικά, διαγραμμικά και μη. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πεδία εφαρμογής, διαφορετικές ρυθμίσεις. Ε, το έχουμε πει πολλές φορές, ε, περιορισμοί διαχωρισμού, ε, των πωλήσεων που γίνονται διαγραμμικά και μη, οι λεγόμενε πωλήσει cross-channel. Κανεί πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να τα ξεχωρίσει. Πού τελειώνει η διαγραμμική, πού αρχίζει η μη διαγραμμική. Ανασφάλεια εννοείται για τον καταναλωτή. Και γι' αυτό πάντοτε προτείναμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογή. Και βεβαίως σημαντικές είναι οι τροπολογίες που εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να επιβεβαιωθούν και από την αξιολόγηση συνεπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συγκεκριμένε τροπολογίες. Χρειάζεται παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα για να μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρουμε. Και επισημαίνω επίσης ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να επισημανθεί ότι με την άρση της οδηγίας του 99 για την προστασία των καταναλωτών δεν προκύπτουν κενά νομικά. Πρέπει να είναι καλυμμένος ο καταναλωτής δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ραγκνέλ. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία τώρα μας έχει δώσει ένα άλλο επίπεδο για το περιεχόμενο μας. Θέλει άλλος το λόγο. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Χάτολα, θέλει κάτι να πει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα θεωρούμε πάρα πολύ θετική την πρόοδο που σημειώθηκε στη δέσμη των νομοθετημάτων για τα ψηφιακά και πρόσφατα εγκρίνεται μία έκθεση σχετική. Έχουμε τώρα τον τριμερή διάλογο, όλα πάνε καλά, επικοδομητικά και ελπίζουμε θα συνεχίσει διαδρομή της η πρόταση. Είπε η κυρία Χαουτάλα ότι και αυτή που, πρόταση που τώρα συζητούμε για τις πωλήσει και αυτή η υπόθεση θα πάει καλά. Βεβαίω είναι αλληλένδετε οι δύο αυτές ε, προτάσει γι' αυτό και εσεί μαζί τα επεξεργάζεστε. Και το Συμβούλιο, όπω είπε η κυρία Χαουτάλα, το Συμβούλιο έχει αρχίσει την συζήτηση και υπάρχει η πρόθεση εξέβραση λύση. άρα είναι και πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο του για την πρόταση αυτή και να καταλήξετε σε μια τοποθέτηση σύντομα. Πολύ ξημών αναφέρεται και θέλω και εγώ να το πω ότι η εμπειρία μας ιδίω όσον αφορά τις ψηφιακές, το ψηφιακό περιεχόμενο μας οδηγεί στο ότι είναι εφικτό να βρούμε κάποια λύση και εμείς επίσης θέλουμε να υπάρξει ευξημένη προσέγγιση για το κάνουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα να μπορούν και οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να κάνουν τις συναλλαγές τους. Άρα χρειάζεται εδώ εξισορρόπηση στη λύση, χρειάζεται ευελιξία. Να τα συζητήσουν και περαιτέρω όποτε χρειάζεται. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Κυρία Χάουταλα, πριν λάβετε το λόγο. Με ενημερώνουν εδώ από τη γραμματεία μας ότι θα είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία για τις τροπολογίες και να πάμε 15 Δεκεμβρίου. Και το κείμενο θα μεταφραστεί κατά την σύνοδο του Στρασβούργου του Ιανουαρίου. Ε, επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η νέα προθεσμή για τις τροπολογίες αφορεί, αφορά συγγνώμη, όχι όλο το θέμα, αλλά μόνο το κείμενο της Επιτροπής και της τροποποίησης της. Ναι, ναι, ναι λέει κύριε Χαρτολά. Ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ, να υπάρξει αυτή η παράταση στην ε, πρόθεσμη αντί για τις 11 του να πάμε παραπέρα. Θα πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις με σκοπό τον συμβιβασμό. Οπότε και προβληματίζομαι γιατί οι συναδέλφοι θα πούνε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί χρειαζόμαστε τα μεταφρασμένα κείμενα. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία τον Ιανουάριο. Δώσαμε αγώνα. Αναβάλαμε την ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ. Πιέζει το χρονοδιάγραμμα για να το καταφέρουμε. Και η κυρία Ρέγνερ είχε μιλήσει γι' αυτό. Τόσο με προβληματίζει αυτό το, το πότε θα έχουμε τις μεταφράσεις. Άρα τι, να μείνει η προθεσμία όπως είχε. Ναι, ναι, ναι, λέει κύριε Χάουταλα. Άρα 5 ώρα στις 11 του μηνός. Ε, για πρακτικούς λόγους. Εκεί καταλήξαμε συμβαστικά. Δεν γίνεται αλλιώ. Θέλετε να μας πει τίποτε άλλο. Ναι, ναι, για το περιεχόμενο. Έχουμε τις μελέτες επιπτώσεις, έχουμε όλα όσα έχει κάνει το Κοινοβούλιο για αυτού του είδους την ε, ε αιώνια η εγγύηση και η πρόταση για τα ψηφιακά όμως δεν λέγει αυτή την ε, ισόβια εγγύηση. Πάντως, εγώ να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό και έτσι όσον αφορά τα υλικά εμπορεύουν τελικά αγαθά να προβλέπεται τέτοια εγγύηση. Έχει να κάνει με την ε, ε, διαρκή ε, τόσο την, την, μακρά ζωή τη διάρκεια αυτών των ε, αγαθών. Άρα, επομένω, κάτι μπορούμε να προβλέψουμε σχετικά σε αυτή την ε, οδηγία. Εσείς κύριε Άγγινερ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ... Όχι, δεν θέλω να πω και το περιεχόμενο, μόνο για τις προθεσμίες. Συμφωνώ με την 11η του μηνός. Είναι ρεαλιστικό να έχουμε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε και καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Χάντολα. Επομένω προτείνει η γραμματεία, λέει ο πρόεδρο, η προθεσμία να οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου στις 7, στις 7. Είναι λίγο σύντομη προθεσμία. Τέλος πάντων, εδώ ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε. Το υπαριθμό 10. Ανταλλαγή απόψεων για την πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι κύριε Χάπροφ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όλη η μέρα δική μου σήμερα. Η Επιτροπή Γιουρία αποφάσισε να εκδώσει μια γνωμοδότηση επί μιας έκθεσης που θα συντάξει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την πολυμορφία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια της ΛΥΜΠΕ είναι η Μπάρμπαρα Σπινέλη από την ΚΟΕ και η Επιτροπή Πολιτισμού και, Εκπαίδευση και Παιδείας αποφάσισε να εκδώσει ως συνδεδεμένη Επιτροπή μια γνωμοδότηση όρισαν τον Κούρτζο Μαλτέζε από την ΚΟΕ ως ε, συντάκτη. Το θέμα αυτό πιστεύω πρέπει να το αναθεωρούμε κάθε λίγα χρόνια διότι παρεμβάλλονται εξελίξεις. Αυτό που συζητάμε εδώ βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοκρατικού κράτους, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η πολυμορφία και η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθούν σημαντικοί πυλώνες που υποστηρίζουν το θεμελιώδης δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης. Αν αποδυναμωθούν αυτοί οι πυλώνες ή αν υπάρχει σχετική ένδειξη, ε, αυτό σημαίνει ότι κάποιος ε, επιχειρεί να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης. Τελευταία έχουμε δει κάποια τέτοια παραδείγματα. Ο συγκλονιστική δολοφονία της ε, δημοσιογράφου στην Μάλτα μας υπενθύμισε αυτό το περιστατικό ότι απειλούνται οι διερευνητικοί δημοσιογράφοι και η προσφέτη έκθεση για τους πληροφοριοδότες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα σε κάποια κράτη μέλη παρατηρούμε συγκέντρωση της εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, με επακολουθεί απειλή ε, της ε, αυτονομίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης να αναφέρω τις ορισμένες ε, χώρες που υπήρξαν ανέκαθεν πολύ ελεύθερες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρατηρούμε κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις. Στη δική μου χώρα, για παράδειγμα, στη Φιλανδία, έγινε μια απόπειρα από επίπεδο Πρωθυπουργού να επηρεαστεί το περιεχόμενο κάποιων νέων υπηρεσιών ε, του, της δημόσιας τηλεοπτικής, τηλεο, ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας ε, και έγινε μια απόπειρα πολιτικού ελέγχου του περιεχομένου και των δημοσιογράφων της ε, κρατικής ραδιοτηλεόρασης, κάτι που αντίκειται στην ελευθερία των μέσων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Εγώ έχω συγκεντρώσει εδώ κάποιες ιδέες για το τι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Πρώτον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εκφράσουμε την ανησυχία μας κατά οποιασδήποτε νομοθετικής προσπάθειας ή διοικητικής προσπάθειας περιορισμού και ελεγχού των μέσων, είτε άμεσα είτε έμεσα. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις περιπτώσεις όπου σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν αρνητικές επιπτώσεις στα μέσα, αλλά οι συνθήκες λειτουργίας τους ε, είναι αυτές που επηρεάστηκαν. Αρχίζοντας να εξετάζω όλες αυτές τις περιπτώσεις, παρατήρησα το ζήτημα της προστασίας των Τον των whistleblower, ε, είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε. Ε, η προστασία δηλαδή των δημοσιογραφικών πηγών. Ως Επιτροπή Αρμόδια για τις περιπτώσεις ε, άρσης ασυλίας ε, συχνά έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις και κατηγορίες της φήμησης. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει μια έκθεση για το θέμα της ελευθερίας των μέσων και έχει πει ότι τα κρατημέλη όπου η δυσφήμιση αποτελεί ποινική, ποινικό αδίκημα θα πρέπει να το αποποινικοποιήσουν. Εδώ και καιρό το ακούμε αυτό και από το Συμβουλίο της Ευρώπης. Επίσης θα ήθελα να αναφέρουμε το ζήτημα των ε, ασφαλών και ε, πολλών διαφορετικών ε, μέσων στα μέσα. Δηλαδή πώς θα ακούγεται η φωνή πολλών μειονοτήτων, είτε μιλάμε για γλωσσικές, είτε για σεξουαλικές, είτε για πολιτικές. Και τέλος, η συγκέντρωση στον τομέα των μέσων. Εκεί δεν θα πρέπει απλά να εξετάζουμε τις κλασικές ε, εταιρείε μέσων μαζική ενημέρωση, αλλά και τα μέσα κοινωνική δικτύωση και άλλε μορφέ μέσων. Εκεί και το ζήτημα των διαφημίσεων ε, όσον αφορά το περιεχόμενο ε, των μέσων κοινωνική δικτύωση και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα της ελευθερίας και τη πολυμορφία των μέσων. Θα ήθελα λοιπόν να, αν θέλετε κάποιοι να μου στείλετε κάποιες ιδέες που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε φυσικά αυτή η γνωμοδότηση θα είναι σύντομη, μια σελίδα. Αυτό δεν μας εμποδίζει από το να κάνουμε και κάποιες τροπολογίες στο σχέδιο κειμένου για να γίνει πιο κατανοητό και πιο πλήρες. Αυτά. Ευχαριστώ. Μίστερ Μαρίνιο Πίντου. Κύριος Μαρίνιο Πίντου. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο και έχω συζητήσει το θέμα αυτό με συναδέλφους ε, ε, στη χώρα μου, άλλους βουλευτές. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Και πραγματική ενημέρωση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει πραγματική ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία του τύπου μπορεί να ασκηθεί κατά τρόπο ακραίο, καταχρηστικό, ε, που να ξεπερνάει το νόημα της ε, εργασίας του ε, δημοσιογράφου, αλλά πάλι πρέπει να διαφυλάσσεται η ελευθερία των δημοσιογράφων που θα πρέπει να είναι σε θέση με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό να παράγει ενημέρωση, πληροφορία προς το συμφέρον της, ε, της κοινή γνώμης των πολιτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα διαμορφώσουν τις θέσεις τους, τη βούλησή τους για να μπορέσουν να διαμορφώσουν πολιτικές θέσεις και επιλογές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορες μορφές εξωτερικής ε, ελευθερία, είτε την εξωτερική προστασία δηλαδή του δημοσιογράφου από την παρέμβαση των λοιπών εξουσιών, πολιτικής, οικονομικής, θρησκευτικής. Όλων αυτών των εξουσιών που βρίσκονται μέσα σε μία κοινωνία και προσπαθούν να ελέγξουν προς όφελός τους ε, τις πληροφορίες ώστε να τους είναι χρήσιμες. Δεν μπορεί ο, δημοσιογράφος λοιπόν να ελέγχεται ή να καθοδηγεί τις τραστοριότητες του από κανένα ή στη δουλειά του από κανένα συμφέρον. Επίσης εσωτερική ελευθερία του δημοσιογράφου και τι εννοώ εδώ. Ε, ελευθερία σε σχέση με την η ιεραρχική δομή μέσα σε μια εφημερίδα, τις αρχές τους προϊσταμένους που μπορεί να τον καθοδηγούν ε, προκειμένου να υπηρετήσει με το έργο του τα οικονομικά ή συνολικά συμφέροντα του ε, εντύπου, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα ε, αντικειμενικά ε, συμφέροντα της ενημέρωσης και επίσης πρέπει αυτή η ελευθερία να είναι ουσιαστική με εγγυήσει που σημαίνουν εγγυήσεις για το δημοσιογράφο, όχι προνόμια, αλλά εγγυήσεις έναντι της κοινωνίας για την ε, πληροφορία που παράγει ένας ε, δημοσιογράφος κατά τρόπο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Και βεβαίως υπάρχουν πτυχές δεοντολογικές, ηθικές. Για το δημοσιογράφο. Όποιος είναι κόλακας, υπηρετεί διαφημιστικούς σκοπούς με την ε, υπόκρυψη σε ειδήσει, προσπαθεί να προσπορήσει όφελος, διαδίδει ψευδείς ειδήσει, πολλαπλασιάζονται οι ψευδείς ειδήσει στο διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν πρέπει να αντισταθούμε σε αυτές τις τάσεις κατάπνιξη της ελευθερίας των ελευθεριών, ένα φαινόμενο που δεν είναι καθόλου καινούριο και καθώς εγώ ε, διατέλασα δημοσιογράφος το αντιπαλεύτηκα αυτό το φαινόμενο πριν από τον Απριλίο του 1974 στην πατρίδα μου την Πορτογαλία επί γράφονταν τόσα ψέματα ότι ήταν ο Μαντέλε ένας επικίνδυνος τρομοκράτης ε, που τον είχαν βάλει στη φυλακή ότι διαδιδόταν η σοσιαλιστική η σταλινιστική προπαγάνδα στην Ευρώπη δεν λεγόταν η, αλήθεια λοιπόν και τα φαινόμενα τα, τα γνωρίζουμε ανέκαθεν Ψευδείς ειδήσει λοιπόν, όπως και παραπλανητική διαφήμιση, είναι στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Ξέρω και εγώ από συνεντεύξεις μου ότι κάπως πρέπει να πω τα πράγματα. Λοιπόν, ε, ας κοιτάξουμε ότι, και ας αναγνωρίσουμε ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιείται το ίντερνετ για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων δεν είναι ε, δεν μπορεί να αποτελέσει μέσον για την περιστολή των ελευθεριών των πραγματικών δημοσιογράφων. Αυτοί πρέπει να δρουν ανεξάρτητα, αυτόνομα, να μην εξαρτώνται από την αυθαιρεσία και την περιστασιακή διάθεση του κάθε προϊστομένου. Και επίσης, μεροληψία το θέμα της μεροληψίας λοιπόν σημαίνει ταυτόχρονα και ένα, ότι μας προσφέρεται ένα μέρος μόνο της ε, αλήθειας. Και μάλιστα υπάρχει το περίφημο ρητό του Μπρέχτ που έλεγε ότι ε, η τυπογραφική μηχανή μπορεί να γράψει πιο πολλά ψέματα από ότι η γράφομηχανή. Ε, σε αυτό πρέπει να σταθούμε, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επανέρχομαι για να πω ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και καλή. Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη θεσμοθετημένη ψευδολογία και πάλι όμως χωρίς ποτέ να αμφισβητούμε ή ακόμα αντίθετα ε, θα πρέπει να ενισχύουμε τα επαγγελματικά, τις επαγγελματικές εγγυήσεις για τον δημοσιογράφο για να έχουμε μια πραγματική και πλουραλιστική ενημέρωση. Thank you, Mrs. Thank you. Η κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Όμως... Μόνο μία σελίδα έχουμε στη διάθεσή μας, άρα πρέπει να είναι πολύ σύντομη η γνωμοδότηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, υποστηρίζω απολύτως τα όσα υπόθηκαν. Ε, ψευδολογία, προστασία, διάψευση μάλλον, προστασία των ε, καταγγελών, των whistleblowers και θα προσέθετα επιπλέον και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων, συνθήκες εργασίας εν γέννη εκείνων οι οποίοι μεριμνούν για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης Πρέπει να γίνουν προσεκτικές έρευνες. Και πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία θέλουμε να αγγίξουμε σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των μέσων κτλ. Αλλά και από την άλλη θα πρέπει να εξασφαλίζεται για τον δημοσιογράφο η δυνατότητα της προσεκτικής επαλήθευσης των πληροφοριών, να μην πιέζεται και χρονικά να γράφει ένα άρθρο, γιατί τότε ε, ε, έρχεται να εμφανιστεί το φαινόμενο της αγέλης ε, στο εντάξει των δημοσιογράφων. Γράφει κάποιος κάτι απρόσεκτα και μετά οι υπόλοιποι τον ακολουθούν, επίσης γιατί δεν έχουν το χρόνο να επαληθεύσουν. Αυτό είναι το ένα. Και πρέπει να διαχωρίσουμε τα fake news από τα false news ψευδείς ειδήσει που σημαίνει αναλυθείς αλλά εσκεμένα ε, και εν γνώση του του είναι αναλυθείς θέμενε στο διαδίκτυο ειδήσει. και μετά υπάρχουν και οι εσφαλμένες ειδήσει που κάποιος αθελά του ενδεχομένως θέτει σε κυκλοφορία. Τα fake news λοιπόν ε, χρησιμοποιούνται, αποτελούν όργανο για την καθοδήγηση της διαδικασίας ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ελευθερία των ΜΜΕ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Τώρα τελευταία για να προστατεύσουμε λέμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πληροφοριοδότες προστασία δηλαδή, των δημοσιογράφων και στην άλλη μεριά το, το, το, το να προστατεύσουμε το δημοσιογραφικό απόρριτο όσον αφορά τι πηγέ. Εάν ένα κράτο δεν μπορεί να κάνει αυτή την προστασία, ε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά την ε, Γαλλία, έχω να σα πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε και στα δύο αυτά μέτωπα. Παρ' όλα αυτά, πέραν αυτού, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει αναδεθεί όπω αναφέρθηκε, είναι η συγκέντρωση των ε, ΜΜΕ σε, στα χέρια των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων οπότε και αυτό έχει μειώσει την πολυφωνία στην ε, Γαλλία ξέσπασε ένα σκάνδαλο πρόσφατα γιατί υπήρχαν κάποια χρηματοδοτικά κέντρα που ανοιχτά είχαν αγοράσει ε, κάποια μέσα και πλήρωναν δημοσιογράφους για να γράφουν αυτά τα οποία συμφέρανε οπότε Έχουμε και τους ε, δημοσιογράφους χωρίς ε, σύνορα που έχουν κάνει κάποια έρευνα και η Γαλλία συνεχώς, συνεχώς κατρακυλάει στη σχετική κατάταξη. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Επίσης σας επισύρω την προσοχή και σε ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται στην ε, Γαλλία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και για άλλες χώρες. Είναι το θέμα του κομφορμισμού Έχουμε δηλαδή κάποιου είδους νόμους που θεσπίζονται όσον αφορά κάποια θέματα που αφορούν την ιστορία της Γαλλίας, παγκόσμια ιστορία της Ευρώπης και που επιβάλλουν συγκεκριμένες απόψεις. Και αν κανείς ε, παρεκκλίνει τότε μπορεί να βρεθεί στο εδόλιο. Και ε, έγινε και κάτι τέτοιο συγκεκριμένα γιατί έγινε μια έρευνα η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την επίσημη ε, άποψη. Οπότε τελικά ε, υπήρχαν διαμαρτυρίες ε, αλλά τέλος πάντων οπότε υπάρχει ένας άλλος νόμος ξέρετε που θεσπίστηκε στη Γαλλία και σύμφωνα με αυτόν υπάρχουν θετικές πλευρές στην απεικιοκρατία. Αυτά λέγανε στο σχολείο. Τα καλά της απεικιοκρατία. και αυτό οδήγησε σε σκάνδαλο, αποσύρθηκε η δημοσίευση, αλλά θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά. Και κατακλείδη να σας πω ότι και εμείς να προσέξουμε, γιατί αφού θέλουμε κείμενα τα οποία καταστήλουν την ρητορική του μίσους, υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος από κάτι, τέτοια φαινόμενα. Προσοχή, έχουμε και την νομολογία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι η ελευθερία έκφρασης αφορά και κάποιες ε, ιδέες οι οποίες σοκάρουν και προβληματίζουν ε, οπότε θα πρέπει να ποινικοποιούμε αλλά να είναι συγκεκριμένο το αντικείμενο όπως η τρομοκρατία ας πούμε αλλά εγώ φοβάμαι από τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις όπως για την ρητορική του μίσους γιατί αυτό είναι πολύ υποκειμενικό να ποιο είναι ο κομφορμισμός από πλευρά του κράτους και αφού μιλάμε για τα fake news προσοχή, προσοχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελευθερία, θα πρέπει να, να η ελευθερία του τύπου και όχι να έχουμε ε, ποινικοποίηση ε, αχαλήνωτη που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σας άκουσα και προβληματίστηκα. Τι θα μπορούσα να συμβουλεύσω την κυρία Χάουταλα, την εισηγήτριά μας, ούτως ώστε να καλύψει και τις δικές μου απόψεις. Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα στην κυρία Χάουταλα. Μα αφού πρέπει να είναι τόσο σύντομη αυτή η έκθεση για ένα τόσο μεγάλο θέμα, τότε έχουμε δύο λύσεις. Ή να ασχοληθούμε το θέμα ουσιαστικά συμβολικά ή αυτή η γνωμοδότηση θα είναι απλά διακοσμητικού χαρακτήρα. Και η Λίμπε θα κάνει την κυρίως δουλειά. Ακριβώς όπως όλοι είπατε, το θέμα αυτό είναι τεραστίας σημασίας. Ε, βέβαια. Και πρέπει να μιλήσουμε για την πολυφωνία, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πολλές επιφυλάξεις για πολλές χώρες, αλλά υπάρχει πολυφωνία. Θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Πάντως αναδύονται κάποια ζητήματα, υπάρχουν κάποιες αρνητικές πλευρές ε, και μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζουν αυτά τα αρνητικά σημεία την λειτουργία των ΜΜΕ. Ναι, λέμε να έχει το κάθε κόμμα, το κάθε κίνημα, την εφημερίδα του, το website του, εντάξει. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό, ναι, να, να ξέρουμε ποιος εκπροσωπεί ποιον. Και ότι εκεί αντικατοπτρίζονται οι απόψεις του τάδε, του, του τάδε κινήματος, του τάδε κόμματος. Και ό,τι έτσι προβάλλονται οι απόψεις. Ναι. Τώρα, πού είναι ο κίνδυνος. Τα ΜΜΕ, τα οποία παρουσιάζουν την αντικειμενική ενημέρωση όταν αυτά περνάνε στο κίνδυνο, στον έλεγχο του κράτους. Θέλει δηλαδή κάποιος υπουργός να παρέμβει για να προβάλλει κάτι. και προβάλλουν αυτά τα ΜΜΕ, ευρεία ενημέρωση, τι απόψει του κόμματο που είναι στην εξουσία. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό και άρα να προσέξουμε σε αυτήν την έκθεση. Είναι κάτι απαράδεκτο. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Η ελευθερία της έκφρασης. Ξέρετε, 20 χρόνια ήμουν δημοσιογράφος και Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα για την ελευθερία της έκφρασης και πάντοτε καταλήγει αυτή η συζήτηση στη διατύπωση κάποιων επιφυλάξεων. Δηλαδή, ποια είναι τα όρια αυτής της ελευθερίας. Είναι η ευθύνη για το τι λέει κανένας. Και συμφωνώ 100% με αυτά που είπε ο κύριος Λεμπρετών. Δεν μπορούμε να πούμε για την ρητορική μίσους στα ΜΜΕ ότι θα πρέπει να αριθμιστεί από την νομοθεσία διότι δεν πρόκειται περί έννοιας ακριβούς. Εάν κάποιος προκαλεί μίσος, ξενοφοβία, ε, ρατσισμό, ε, αν κάποιος καταφέρεται κατά άλλων θρησκειών, τι θα κάνουμε θα δεχθούμε μια τέτοια στάση. Δεν είναι καταδικαστέα. Το θέμα είναι η ευθύνη για τους λόγους εκάστου. Πολλές φορές επομένως μια τέτοια συμπεριφορά επιδέχεται ποινική δίωξη. Αυτό έχω να σας πω ως δημοσιογράφος. Αν θέλουμε οι δημοσιογράφοι να λειτουργούν σε καλές συνθήκες και με ελευθερία αυτό είναι δύσκολο. Ναι, ναι, ναι, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω, του λέει ο πρόεδρος να ε, ολοκληρώσει του ομιλητού. Οπότε γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατοχυρώσουμε αυτή την δημοσιογραφική ελευθερία, γιατί οι δημοσιογράφοι γενικώ ε, υφίστανται κάποια επιρροή από τους προσταμένους τους, ε, από το, το κοινό τους, από τους, τους πελάτες τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Όμω έχουν την υποχρέωση οι δημοσιογράφοι να επαληθεύουν κάθε πληροφορία που του δίνεται ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω και εγώ δύο σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά σχετίζονται με το ζήτημα της ασφάλειας. Διότι το ψέμα αποτελεί πλέον επίσημο όπλο του Κρεμλίνου το χρησιμοποιεί για την προπαγάνδα του, για το στρατιωτικό του δόγμα. Το δόγμα Γερασίμοφ χρησιμοποιεί διαφάνειες. Ε, οπότε έτσι πρέπει να το δούμε. Πρέπει να υπάρχει ευθύνη. Όχι να μιλάμε μόνο για την ελευθερία των μέσων, αλλά και για την ευθύνη των μέσων. Αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Και η τρίτη μου παρατήρηση. Δεν κατάλαβα τι είπαν ο κ. Μανώκη για την Σοβιετική Ένωση γιατί στη μετάφραση μου είπαν ε, ότι είναι ψευδής είδηση το ότι η Σοβιετική Ένωση έχει πράκτορα στην Ευρώπη. Ίσως να υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση διότι ένας από τους πράκτορες ε, ε, από τη Γερμανία τώρα ε, υπήρξε με την Ρωσική Ομοσπονδία πρόεδρε, για ένα διάστημα, ξέρετε, ε, κατέκλυζαν την Ευρώπη ψευδείς ειδήσει από την Σοβιετική Ένωση. Οπότε σήμερα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό των ψευδών ειδήσεων. Είναι κάτι φυσικό το οποίο σχετίζεται με την ελευθερία του τύπου.